Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι έχετε λάβει το χνοδιάγραμμα των συνεδριάσεων για φέτος, από κοινού και με το σχέδιο ημέρησης διάταξης. Ξέρετε ότι η Επιτροπή Ήτρα καλύπτει όλες ε, τις γλώσσες. Τα έγγραφα δεν μπορείτε να τα βρείτε τυπωμένα, μόνο στο διαδίκτυο στο πλαίσιο της διαδικασίας paperless. Ευχαριστώ την ε, γραμματεία που προετοίμασε αυτό το πακέτο υποδοχής που σας ε, μοιράστηκε την περασμένη εβδομάδα. Το θεώρησα πολύ ενδιαφέρον και ε, βοηθάει τα νέα μέλη να εξοικειωθεί με το περιεχόμενο της Επιτροπής μας. Μπορείτε να το βρείτε και στον ιστότοπό μας βέβαια. Όσοι ήθιστε, μεταδίδετε και μέσω διαδικτύου συνεδρίασή μας σε 21 γλώσσες. Στο φάκελό σας έχετε και τα πρακτικά της 10ης Ιουλίου. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, θα εγκριθούν. Επόμενο σημείο στη μεσαδιάταξη είναι ο Γενικό Προπολογισμό Ευρωπαϊκή Ένωση για, την για, την, ε, για το οικονομικό έτος 2020, όλα τα τμήματα. Συμφωνήθηκε με τους ε, συντονιστές την περασμένη φορά να καταρτήσω ε, την γνωμοδότηση, την οποία θα σας παρουσιάσω τώρα εν ολίγης. Η Επιτροπή λοιπόν κατέρτισε τον προπολογισμό, το σχέδιο προπολογισμού για το 2020 στις αρχές Ιουνίου. Πρότεινε να συμπεριλάβει ε, πιστώσεις ανάληψης δεσμεύσεων στον ε, τίτλο 1α κατά 5,5% και ε, πιστώσεις πληρωμή κατά 7,7%. Όμως ε, η Επιτροπή παραμένει κάτω από το όριο του τίτλου 1α κατά 474,6 εκατομμύρια ευρώ. Και πάλι λοιπόν η Επιτροπή είναι ήδη κάτω από το όριο. Μετά, στις αρχές Ιουλίου, το Συμβούλιο αποφάσισε επί της θέσης του και ε, περιέκοψε περαιτέρω το 1α κατά 747,4 εκατομμύρια. Περαιτέρω λοιπόν περικοπές και από το Συμβούλιο σε σχέση με την πρόταση τη Επιτροπή. Το σχέδιο γνωμοδότησή μου, λοιπόν, προτείνω να αξιοποιήσουμε όλο το περιθώριο που έχουμε στο 1α και να αξιοποιήσουμε το μηχανισμό ευελιξία, καθώ ε, ε, Κενέ διατάξει του χρηματοδοτικού κανονισμού που επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση των ε, ε, πιστώσεων για τον τομέα της έρευνας και μόνο. Προτείνω λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα. Δεν σημαίνει αυτό βέβαια ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σύνολο του περιθωρίου ε, σε συγκεκριμένου τομεί, γιατί υπάρχουν και άλλοι όπω ε, η εκπαίδευση, οι μεταφορέ, που επίση περιλαμβάνονται στον τίτλο του προπολογισμού αυτού. Πρέπει λοιπόν να εξευρεθεί μια ισορροπία μεταξύ των επιμέρου ε, τομέων πολιτική. Προτείνω αυτή την άγουσα για το 2020 είναι και η τελευταία χρονιά του τρέχοντο ΠΔΠ. Γι' αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε ως μια γέφυρα προς το επόμενο ΠΔΠ γιατί από την εμπειρία μας βλέπουμε ότι σε ένα νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, ξεκινάμε συνήθως αργά. Γι' αυτό είναι καλό να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο τους διαθέσιμους πόρους για την ε, χρονιά που έρχεται. Επιπροσθέτως, έχουμε δύο σημαντικά προγράμματα, το Horizon 2020 και το COSME, για το οποίο έχουμε ξεπεράσει ε, τα όρια. Αυτά τα προγράμματα λοιπόν μπορούν εύκολα να αξιοποιήσουν περισσότερους ε, πόρους. Αναφέρθηκα στις περικοπές του Συμβουλίου που έχουν να κάνουν με το κοινό στρατηγικό σχέδιο πλαίσιο για την έρευνα και καινοτομία, 429,9 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 430 αφορούν το πρόγραμμα Horizon 2020. Η μηχανισμός συνδέονται στην Ευρώπη, 197 εκατομμύρια, εκ των οποίων 169 αφορούν τις μεταφορές και 28 ε, την τεχνολογία της πληροφορίας. GFC, μείον 90 εκατομμύρια και ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κόσμε, Εκεί η περικοπή ήταν κατά 20 εκατομμύρια. Θα ήθελα λοιπόν να επισημάνω προς τους νέους συναδέλφους ΣΥΤΡΕ ότι πάντα το ίδιο ακούμε από το Συμβούλιο, όπως και σήμερα το πρωί από την Προεδρία. Πόσο σημαντική είναι η έρευνα, η καινοτομία και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά μετά όταν πρέπει να μιλήσουν οι πράξεις και όχι τα λόγια, το Συμβούλιο τα αλλάζει. Δεν ακολουθεί τις ίδιες προτεραιότητες, αλλά προχωρά σε περικοπές. Επί τη πρόταση τη Κομισιόν δεν μπορούμε να δεχθούμε κάτι τέτοιο, γι' αυτό θα καταθέσω τροπολογίε για την ε, αναστολή όλων των περικοπών που έχει προτείνει το Συμβούλιο. Μετά έχουμε και το θέμα των ε, ευρωπαϊκών οργανισμών ε, στο δικό μα πεδίο δραστηριοποίηση, γιατί παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των πολιτικών. Χρειάζονται λοιπόν και τους απαραίτητους πόρους ε, και μέλη προσωπικού για να μπορέσουν να επιτελέσουν το έργο τους. Και κάθε χρόνο βλέπουμε ότι αυξάνονται οι πολιτικές, αυξάνεται το, ο φόρτος εργασίας και γι' αυτό πρέπει να τους δώσουμε και τα αντίστοιχα κονδύλια για να μπορέσουν να προσλάβουν εμπειρογνώμονες και να επιτελέσουν το έργο τους, αυτά τα νέα καθήκοντα. Πιο συγκεκριμένα για τον Acer. Για την ενέργεια, λοιπόν, εδώ βλέπουμε υποχρηματοδότηση εδώ και χρόνια και μέσω της νομοθεσίας που υιοθετήθηκε κατά την τελευταία θητεία, ο οργανισμός αυτός αποκτά ακόμα νέες δραστηριότητες και αρμοδιότητες. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να αυξηθεί το προσωπικό και η χρηματοδότηση για τον Acer. Και εδώ θα καταθέσω κάποιες ε, τροπολογίες για να εισαγάγουμε γραμμέ προπολογισμού πάνω από τα επίπεδα που προτείνει η Κομισιόν. αλλά και σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες ε, της Ήτρε, όπως ε, ο ορίζον και το ΣΕΦ ε, για την ενέργεια. Αυτά έχω κάνει μέχρι τώρα. Με ενδιαφέρον περιμένω και τις δικές σας τροπολογίες και σίγουρα θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε επί ενό ε, καλού πακέτου που θα ωφελήσει ε, και τον κλάδο, τη βιομηχανία ε, και τους οργανισμούς και τους πολίτες. Λοιπόν, έχουμε δύο προθεσμίες για τις τροπολογίες. Αύριο, σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες επί του προϋπολογισμού και η άλλη προθεσμία λίγη στις 3 Σεπτεμβρίου. 5 Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό είναι η προέδρο. Ωραία. Αυτά είναι ολίγη ε, από εμένα. Εάν έχετε ερωτήσει, είμαι στη διάθεσή σα και βεβαίω μπορούμε να ακούσουμε και προτάσει που σίγουρα θα έχετε. Ποιος θα να πάρει το λόγο. Η κυρία Σπυράκη πρώτη. Για άλλη μια φορά, ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Απλά ήθελα να πω ότι μας παρουσιάσετε ε, μια εμβριθή μελέτη και θα ήθελα να επισημάνω κάποια θέματα που είναι πολύ σημαντικά. Καταρχήν, όσον αφορά ε, τα προγράμματα Horizon και COSME, συμφωνώ ότι πρέπει να έχουμε ένα πιο φιλόδοξο προπλογισμό για το 2020 ε, Βεβαίω δεν θα πρέπει να υποχρηματοδοτούνται προγράμματα, πρέπει να στηρίξουμε τα πανεπιστήμια μας, ε, τους ερευνητικούς φορείς, ε, τις επιχειρήσεις μας. Όσον αφορά την πλήρη οικονομική υποστήριξη προς τους ε, οργανισμούς που εμπίπτουν στη δική μας τα αρμοδιότητα, όπως είναι ο ΕΝΙΖΑ, πιστεύω ότι ο ΕΝΙΖΑ θα δραματίσει καθοριστικό ρόλο στα θέματα κυβερνοασφάλειας και γι' αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξει περαιτέρω χρηματοδότηση του φορέα ΕΝΙΖΑ. Και χρειαζόμαστε όχι μόνο επιπρόσθετα κονδύλια για να καλύψουμε τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των Συμφωνίας των Παρισίων, αλλά πρέπει να έχουμε και περισσότερα κονδύλια για μεταβατική περίοδο, για περιοχές που εξαρτώνται ε, πολύ από τον άνθρακα. Αυτό πρέπει να αναφέρεται στην γνωμοδότησή μας, γιατί είμαστε Επιτροπή Βιομηχανίας και η κυρία Φοντελάιν ανέφερε ήδη ότι θα υπάρξει επιπλέον χρηματοδότηση για περιοχές που εξαρτώνται από τον άνθρακα. Και τέλος, ε, ε, θέλω να απογραμμίσω ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η χρηματοδότηση για την ε, Interconnecting Europe Facility και άλλη μια φορά λοιπόν σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γκάια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που θα συνεργαστούμε και στο σημείο αυτό θέλω να σας πω ότι είμαι ο σκιώδης εισηγητής των σοσιαλδημοκρατών για αυτό το θέμα. Και βασικά θέλω να σας πω ότι έφυγα από την Επιτροπή Προπολογισμού ε, και πέρασα στην Επιτροπή Βιομηχανίας ε, για να ασχοληθώ με τα νομοθετικά. Αλλά ε, παρόλα αυτά, επειδή εδώ πρόκειται για θέματα προπολογισμού, πολύ ευχαρίστω θα ασχοληθώ. Τα ξέρω τα θέματα προπολογισμού και γι' αυτό η ενασχόλησή μου θα μου προκαλέσει και ευχαρίστηση. Αναφερθήκατε ένα περικοπέ σε αυτό τον τομέα. Το Συμβούλιο το κάνει αυτό πάντα με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Εγώ όμω εδώ θέλω να επισημάνω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα 474,6 εκατομμύρια ευρώ είναι κάτω από το όριο ε, το οποίο θα οριζέ το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Άρα υπάρχει περιθώριο προς τα επάνω για να μπορέσουμε να επιτύχουμε ευξήσει. Ε, ίσως το Συμβούλιο να μην χαρεί, αλλά στη τελική ανάλυση αν δεν υπάρχει και αυτή η ένταση ε, δεν χαίρεται κανείς και όλα στις διαπραγματεύσεις. Ο συνήθως το Συμβούλιο έκανε περικοπές και αυτό που με πικραίνει λιγάκι είναι ότι πλήττονται προγράμματα των οποίων η σημασία κατ' ουσίαν αναγνωρίζεται από όλες τις πλευρές και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Connecting Europe Facility, Horizon, Cosme, αυτά θα πληγούν. Και γι' αυτό εγώ υποστηρίζω ανεπιφύλακτα ε, το να αυξηθούν αυτές οι γραμμές του προπολογισμού που έχουν περικοπεί. Και πέρα από αυτό θα καταθέσω και κάποιες άλλες τροπολογίες. Κατά την προηγούμενη θητεία σε όλες τις διαδικασίες προπολογισμού ε, επιλέξαμε εκείνες τις ε, γραμμές ε, για στρατηγικές επενδύσεις που είχαν περικοπεί και αυτές ε, επανήλθαν στο αρχικό τους ύψος για να καταστήσουμε σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό το νέο εργαλείο, το ΕΦΣΥ, ναι μεν το χαιρετίζει, αλλά θα ήθελε το ποσό της εγγύησης που πρέπει να εφίσταται, να χρηματοδοτείται από φρέσκα λεφτά των κρατών μελών και όχι να χρηματοδοτείται από ποσά που θα έχουν περικοπεί από άλλες γραμμές. Ε, εγώ αυτή είναι η γραμμή που θέλω να ακολουθηθεί και νομίζω ότι συμφωνούμε ε, πρόκειται για επαρκή χρηματοδότηση για το προσωπικό που θα εργαστεί στους ε, οργανισμούς. Ε, εμείς συμφωνούμε με αυτό. Ενίζα, ΕΣΑ, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας, όλοι αυτοί οι οργανισμοί, αλλά και άλλοι έχουν ανάγκες. Αυτοί οι οργανισμοί πρέπει να λειτουργούν. Ακούσαμε γιατί. Βλέπουμε όμως να προκύπτει επανειλημμένα μια κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι πρόθυμη να διαθέτει απαραίτητα κονδύλια για αυτούς τους οργανισμούς. Εγώ στην Επιτροπή Προϋπολογισμού είχα συνηθίσει να μην αντιδρώ καν στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά να αντιδρώ στα αιτήματα των οργανισμών. Γιατί έχω κάνει την εμπειρία ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει κάνει πολύ μεγάλες άδικες περικοπές στους οργανισμούς. Γι' αυτό λοιπόν ε, εγώ θα ξεπερνούσα όπου μπορεί κανείς βέβαια ε, την πρόταση της Επιτροπής, κλιματικές αλλαγές, συμμετοχή σε μία κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, εκεί εγώ ενδεικτικά θα, αύξ, θα, θα προτιμούσα να υπάρχει αύξηση των κονδυλίων. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Η κυρία ε, Νταμπάουβα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ είμαι σκιώδης ε, της ε, ομάδας μας ε, και όπως και ο κύριος Γκάιερ και εγώ ασχολούμαι με τον προϋπολογισμό εδώ και αρκετό καιρό από διαφορετικό πρίσμα ασχολούμαι στον έλεγχο προϋπολογισμών για την αποτελεσματικότητα των δαπανών. Η δική μου πολιτική ομάδα πιστεύει ακράταντα ότι έχουμε ε, δαπάνες για την έρευνα και την καινοτομία και αυτές είναι απολύτως απαραίτητες για να ε, ικανοποιήσουμε τους στόχους του κλίματος. Άρα δηλαδή είμαστε υπέρ της αύξησης της χρηματοδότησης το 1α και ε, θέλουμε να είμαστε και πιο φιλόδοξοι για την καθαρή τεχνολογία. Άρα δηλαδή να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο της ευελιξίας όπως πολύ σωστά είπατε. Παράλληλα, όπως ακριβώς αναφέρθηκε, είναι απολύτως απαραίτητο οι οργανισμοί να χρηματοδοτούνται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Δεν μπορούμε να τους φορτώνουμε νέες αρμοδιότητες χωρίς να τους προσφέρουμε και τα απαραίτητα κονδύλια. Και αυτό ισχύει κυρίως για τον, τον φορέα ένση και άλλους. Ε, τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οι νέες πρωτοβουλίες δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται απαραίτητα από τη μείωση άλλων, μείωση άλλων προγραμμάτων. Ευχαριστώ που συντάξατε αυτή την γνωμοδότηση και με μεγάλη μου χαρά θα συνεργαστώ μαζί σας. Thank you. Ε, Mr. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Νινιστό Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ήταν πολύ καλή βάση η παρουσίασή σας. Ε, να συμπληρώσω μόνο ότι οι δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα δυστυχώς ε, δεν είναι αρκετές στο σχέδιο προπολογισμού. Ιδίως αν δούμε το πρόγραμμα Horizon 2020 για την επταετία το κλίμα είναι 26,44%. Ε, θα πρέπει να είναι 35%. Είμαστε πολύ κάτω λοιπόν από το στόχο. Θα μπορούσε να ε, βελτιωθεί η χρηματοδότηση σε ό,τι αφορά λοιπόν τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων. Θα πρέπει να, να εξετάσουμε αυτό το τομέα σε σχέση και με το κλίμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν μπόρεσα να ακούσω πλήρω την παρέμβασή σα, Πρόεδρε, γιατί χρειάστηκε να απαντήσω ένα τηλέφωνο. Συμφωνώ απόλυτα με την παρέμβαση του αδέλφου Γκάιερ, όπω και άλλε συνάδελφοι, γιατί πιστεύω ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή από την Επιτροπή μια μείωση κεφαλαίων που ανταποκρίνονται σε προγράμματα που μετά όλοι, το Συμβούλιο, η Επιτροπή, έρχονται και μας λένε ότι είναι θέματα προτεραιότητας. Αν είναι προτεραιότητας, να χρηματοδοτηθούν κατάλληλα. Αλλιώ δεν μπορεί να ανεχθούμε τέτοιες ανισότητες. Κατόπιν, αυτό που είναι σημαντικό είναι οι περικοπές οράζων και κόστλε μικρά, μικρές περικοπές, αλλά σημαντικές. Όλοι μιλάμε για διεθνοποίηση, ψηφιοποίηση, κατάρτιση κλπ. Κατάρτιση προσωπικού για να αντιμετωπιστούν τις αλλαγές. Ο, εγώ συμφωνώ λοιπόν απόλυτα με την εισηγήτρια και τους σκιώδεις που ζητούν την αποκατάσταση ε, των κονδυλίων σε επίπεδα ελάχιστα ε, κατ' ελάχιστον αποδεκτά. Πρέπει να προκαλέσουμε και το Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Για τις υπηρεσίες τώρα, πιστεύω ότι κάποιες από τις υπηρεσίες χρειάζονται μία προσαρμογή της χρηματοδότησής τους και του προσωπικού. Όχι όλες. Θα πρέπει να κάνουμε μία πιο επιλεκτική προσέγγιση. Άσερ, για παράδειγμα, παίρνει αρμοδιότητες συνεχώς χωρίς να έχει αύξηση του προσωπικού της. Και άλλες υπηρεσίες χρειάζονται αύξηση του προσωπικού κατά πασφαιρότητα. Αυτό όμως δεν μπορούμε να το κάνουμε γενικά, οριζόντια και αδιάκριτα για όλες. Επανέρχομαι στα βασικά. Δεν μπορούμε να δεχθούμε μία μείωση. Προτείνω να αποκαταστήσουμε τις αρχικές, ε, τα αρχικά ποσά και να παρακολουθήσουμε τι θα γίνει στην ε, Επιτροπή Προπολογισμών και στην Ολομέλεια, ζητώντας να τηρηθούν οι δικές μας επιλογές γιατί είναι απλά ρεαλιστικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καταρχά, πρέπει να δούμε ότι στη φάση αυτή είναι δύσκολο να αυξήσουμε τα κονδύλια. Αλλά ταυτόχρονα δεν μπορείτε να γνωρίσετε ότι φεύγει ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες της Ένωσης. Ζητάτε και άλλη χρηματοδότηση για το Horizon 2020. Πώς θα γίνει κάτι τέτοιο όταν όλες οι επιτροπές ζητούν αύξηση. Τέλο πάντων, εσεί θα το πληρώσετε, όχι εγώ. Αν θέλετε να σα δουν σοβαρά, πρέπει να αναγνωρίσετε ποια είναι η πραγματικότητα και να αντιμετωπίσετε την πραγματικότητα όπω έχει. Κυρία Καρβάλιο. Ευχαριστώ. Υποστηρίζουμε απόλυτα το έργο σας, το σχέδιο γνωμοδότησης και την αναστροφή των περικοπών σε προγράμματα που είναι τόσο σημαντικά για την οικονομική ευημερία και ανάπτυξη των πολιτών μας. Τρία θέματα θέλω να υπογραμμίσω. Είπατε το τεράστιο να αύξει την υπερβολική συμμετοχή στο Horizon 2020, την ανάγκη συμμετοχής κάποιων κρατών που έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή στο Horizon 2020 και στο κόσμο. Να τονίσω τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατή ευελιξία και την επαναχρησιμοποίηση των πόρων της Επιτροπής για την έρευνα, να το αυτή τη, να τονίσουμε αυτή τη δυνατότητα και την έμφαση στις καθαρές τεχνολογίες αλλά και στην τεχνολογία της πληροφορικής. Ευχαριστώ και έχετε την υποστήριξή μας. Ο κ. Γεωργίου. Της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς θα καταθέσουμε διάφορες τροπολογίες προτείνοντας ανακατανομή των κοντιλίων με στόχο να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι ανάγκε τη κοινωνία, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τη ραχοκαγιά τη οικονομία μα, αλλά και τη βιομηχανία, ιδιαίτερα των κρατών μελών που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση. Μια τέτοια χώρα είναι και η δική μου, η Κύπρο. Κατά την άποψή μα, η πρόταση τη Κομισιόν για αύξηση των επενδύσεων στην αμυντική βιομηχανία με στόχο την περαιτέρω στρατιωτικοποίηση τη Ένωση αποτελεί μια αρνητική εξέλιξη. Με τροπολογία λοιπόν θα ζητήσουμε το κοντήλι των 255 εκατομμυρίων, το οποίο προορίζεται για τι πολεμικέ βιομηχανίε, να δοθεί στο πρόγραμμα COSME καθώ και στο πρόγραμμα Ορίζοντα 2020, ώστε να αξιοποιηθεί για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα ζητάμε να αυξηθεί το ποσό που δίνεται για βελτίωση τη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, καθώ και το κοντήλι για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω τη έρευνα και τη καινοτομία με στόχο τη δημιουργία νέων αξιοπρεπών θέσεων εργασία. Εξίσου σημαντική είναι και η τροπολογία που έχουμε καταθέσει προτείνοντα να αυξηθεί το κοντήλι για αποτελεσματική αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή. Έχουν λεχθεί πολλά για αυτό το πράγμα. Θα επανέλθουμε σε βάθο πιο ύστερα. Ε, επιπλέον, αναφέρομαι σε μια πολύ σημαντική τροπολογία που έχουμε καταθέσει μαζί με ευρωβουλευτές διάφορων πολιτικών ομάδων για τη δημιουργία ενός πιλωτικού προγράμματος για την αντιμετώπιση του παιδιατρικού καρκίνου. 6.000 παιδιά και νέοι πεθαίνουν κάθε χρόνο στην Ευρώπη από καρκίνο. Έχουμε χρέος και καθήκον ως άνθρωποι να σταματήσουμε αυτήν την μάστιγα. Προτείνουμε λοιπόν να δημιουργηθεί αυτό το πρόγραμμα το οποίο θα αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη και με συλλογική προσπάθεια να βελτιώσουμε τις διαδικασίες διάγνωσης της νόσου και ιδιαίτερα την ανάπτυξη νέων αποτελεσματικών θεραπείων. Ευχαριστώ. Thank you Κάποιος άλλος ε, παρακαλώ, ε, αν όχι θα ήθελα να δώσω, θα έδινα το, ρόλο στην, το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, θα ήθελα να πω εγώ το εξή. Επισημάνατε, κατά την άποψή μου, διάφορες καταστάσεις Έγινε λόγος ε, για το πρόγραμμα της, ε, για το Ταμείο της ε, Δίκαιης Μετάβασης. Γνωρίζουμε ότι στο Ταμείο αυτό θα υπάρχουν φρέσκα χρήματα και όχι κονδύλια που θα έχουν περικοπεί από άλλες γραμμές. Αυτή είναι η γραμμή και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο ε, για τα προγράμματα για τα οποία είμαστε αρμόδιοι. Επίσης, όταν μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες στους ε, οργανισμούς, ε, θα πρέπει να μεταφέρουμε και προπλογισμούς, αλλιώς όλο αυτό το θέμα δεν θα λειτουργήσει. Ευελιξία για την έρευνα, όλα αυτά είναι πολύ καλές ιδέες. Προσβλέπω στις τροπολογίες σας και να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει κάποια ημερομηνία, αν δεν τις έχετε καταθέσει όλες, τον Σεπτέμβριο. On the budgetary amendments on 3rd of September, yes, to make sure we can. um, so the budgetary amendments we need to vote on. Για τις τροπολογίες ε, θα πρέπει, για τον προβλησμό θα πρέπει να ψηφιστούν μέχρι τις 3 ε, Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό ε, υπάρχει αύριο η καταληκτική ημερομηνία για τα υπόλοιπα. Θα ψηφιστούν 5 Σεπτεμβρίου και κατά τα άλλα θα σας τα πω στην επόμενη συνεδρία. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το θέμα στην ημερήσια διάταξη και τώρα μπορούμε να καλέσουμε τον πρώτο καλεσμένο για σήμερα το απόγευμα από τους φορείς, τον κύριο Ποτότσνικ, ο οποίος είναι διευθυντής του φορέα Acer. Uh, uh, uh, well, Καλώς ήρθατε, κύριε Ποτότσνικ. Βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας θητείας. Θεωρήσουμε λοιπόν καλό ήδη να προσκαλέσουμε τους εκπροσώπους ε, των ευρωπαϊκών οργανισμών με ιδιαίτερη έμφαση στον ACER Μπορείτε λοιπόν στην συντομία να μας ε, παρουσιάσετε τον φορέα σας, ε, την κατάσταση σήμερα και άλλα θέματα που σας ε, αφορούν και σας ενδιαφέρουν. Παρακαλώ. Μετά θα ακούσουμε και τους συναδέλφους, τους ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ήτρε. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να σας απευθύνω το λόγο τόσο νωρίς στη θητεία σας και σας ευχαριστώ πολύ και για τα πολύ καλά σας λόγια προηγουμένως, το προηγούμενο θέμα της μεσαιδιάταξης Διάταξης όπου στηρίξατε τον Acer τα οποία ισχύουν, γιατί και εμάς μας προβληματίζει. Βλέπουμε ότι αναλαμβάνουμε όλο ένα και περισσότερες αρμοδιότητες και αυτό είναι πολύ θετικό βέβαια, χωρίς όμως να βλέπουμε μια αντίστοιχη αύξηση των πόρων μας. Και πραγματικά καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτελέσουμε το έργο μας εδώ και πολλά χρόνια και θα σας τα παρουσιάσω και στη συνέχεια. Έχει διανεμηθεί υλικό προς εσάς, δεν ε, θέλω να τα παρουσιάσω όλα διεξοδικά, περισσότερο προς ενημέρωσή σας είναι. Υπάρχουν όμως και στοιχεία που δεν θα καλύψω στη σημερινή παρουσίαση, ίσως ε, καλυφθούν στη συνέχεια στις ερωταπαντήσεις, άμα σας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, ο φορέας ιδρύθηκε στο πλαίσιο της τρίτης δέσμης ε, για την ενέργεια, όπου δημιουργήθηκε ένα νέο ε, θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο, και από πλευρά κανονιστικού πλαισίου και από πλευρά συστήματο έπρεπε να δημιουργηθεί νέο φορέα και από πλευρά ρυθμιστική αρχή είναι ο Acer αυτό που το έχει αναλάβει αυτό το έργο. Θα σα παρουσιάσω λοιπόν τον ρόλο του οργανισμού έως τώρα. Πώ θα αλλάξει αυτό ο ρόλο με τη δέσμη καθαρή ενέργεια που θα τέθει σε ισχύ, όπω γνωρίζετε καθώ εσεί το υιοθετήσατε, Πώ συμβάλλουμε εμείς στην επίτευξη των στόχων για τους Ευρωπαίου καταναλωτές ε, και η μόνιμη δημοσιονομική μας κατάσταση. Το 2011 δημιουργήθηκε λοιπόν ο Acer στο πλαίσιο της ε, ολοκλήρωσης της ενιαία αγοράς. Και εμείς θεωρούμε ότι προωθούμε ε, τρεις φορείς, ό,τι αφορά την, ε, τρεις τομείς μάλλον, την ολοκλήρωση της αγοράς, ε, την ανάπτυξη υποδομών, αλλά και την ε, εποπτεία της αγοράς. που είναι πολύ σημαντικά και από πλευρά ασφάλειας εφοδιασμού. Ιδιαίτερα η εποπτεία της αγοράς είναι κάτι που αναλάβαμε εμείς μετά την ίδρυσή μας, αλλά γίνεται όλο ένα και πιο σημαντικό στοιχείο προκειμένου η ενέργεια να ε, την χάνει εμπορία σε σύμφωνα με τα καλύτερα δυνατά πρότυπα. Ο οργανισμός λοιπόν βασίζεται σε εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις προς ε, ε, τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, τους παρόχους και τα ευρωπαϊκά δίκτυα και τα θεσμικά όργανα. Μέχρι τώρα είχε την αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις μόνο σε ειδικέ ε, περιπτώσεις. Όταν δηλαδή οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν μπορούσαν να αποφανθούν ή αποφάσιζαν να μεταβιβάσουν ε, την ευθύνη και την αρμοδιότητα προς ε, τον οργανισμό. Εδώ έχετε έναν πιο διεξοδικό κατάλογο, όχι πλήρη βέβαια, των καθηκόντων μας. Στους τρεις φορείς που σας, μη, συγγνώμη, που προανέφερα. Δεν θέλω να επισέλθω σε όλους αυτούς, μπορούσα να το κάνω στη συνέχεια αν το θέλετε. Μία πτυχή μόνο να επισημάνω, την παρακολούθηση της αγοράς, που είναι πολύ βασικό μέλημα της ε, υπηρεσίας μας. Παλιότερα εστιάζαμε περισσότερο στην ανάπτυξη της αγοράς, αλλά τώρα έχουμε να κάνουμε και με τους κωδικούς δικτύων, σε ό,τι αφορά του ε, συγκεκριμένου κανόνες που έχουν να κάνουν με την αγορά και τα συστήματα. Μέσω λοιπόν τη ε, παρακολούθηση της αγοράς που ε, εκπονεί ο Acer και έχουμε εκθέσεις κάθε χρόνο, ελπίζω να καταφέρουμε να την παρουσιάσουμε και στην Επιτροπή σας. Εκεί λοιπόν επισημαίνουμε τι θα μπορούσε να βελτιωθεί, αλλά και τι βαίνει καλώς στην ευρωπαϊκή αγορά. Θα ήθελα λοιπόν εν συντομία να σας δείξω ορισμένα από τα αποτελέσματα των ε, δραστηριοτήτων μας ε, στον τομέα παρακολούθησης αγοράς. Όπως ξέρετε, ε, στην Day Ahead Market έχουμε σχεδόν πλήρω συνδεδεμένη αγορά. Εκεί λοιπόν η ηλεκτρική ενέργεια τυχάνει εμπορία χωρί προσκόμματα. Έχουμε λοιπόν τον μπλε τομέα δυτικά και νότια και σε κόκκινο βλέπετε την αγορά 4M. Με την ε, σύνδεση της αγοράς λοιπόν έχουμε σημαντική ωφέλεια σε ό,τι αφορά την ε, διασυνοριακή ικανότητα. Εδώ λοιπόν εκτιμούμε τα επίπεδα αποδοτικότητας σε ό,τι αφορά τους διασυνοριακούς ε, τομή διασύνδεσης ε, όταν όλα αυτά αξιοποιούνται σωστά. Από το 2012 μέχρι το 2014, λοιπόν, τα βλέπετε αυτά, όταν υπήρξε η σύνδεση της αγοράς, ε, η αποδοτικότητα βελτιώθηκε από το 60% στο 85%. Όλα αυτά ωφελούν τελικά τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Και στη τελική ανάλυση μόνο έτσι μπορούμε να αξιολογήσουμε το έργο μας. Ε, εκτιμούμε κατά πόσο βελτιώνει την ε, καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Και βλέπουμε ότι αυτό συμβαίνει. Δεν έχει ολοκληρωθεί βεβαίω το έργο μας. Κάποιες φορές βλέπουμε ότι η ηλεκτρική ενέργεια κατευθύνεται, ε, ακολουθείται λάθος κατεύθυνση. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ποσό τη τάξη των 200-250 εκατομμυρίων ε, κάθε χρόνο. Η ολοκλήρωση λοιπόν τη ε, σύνδεση αγορά είναι πολύ σημαντικό ε, στόχο. Βέβαια, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και σε άλλους τομείς, και στο intraday και στο balancing. Τώρα, τα τελευταία 3-4 χρόνια βλέπουμε, από τότε που αρχίσαμε να εντοπίζουμε το πρόβλημα το 2015 και το 2016. Καταρτήσαμε μία ε, σύσταση και είδαμε με τα χαρά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την συμπεριέλαβε στην δέσμη για την καθαρή ενέργεια. Αναφέρθηκα λοιπόν στην ε, χρήση των interconnectors και την ικανότητά τους και τώρα πρέπει να δούμε τι, πόση ικανότητα παρέχεται στην αγορά. Και εμείς εκτιμούμε ότι θα μπορούσε να δοθεί μεγαλύτερη ικανότητα στους διασυνορικούς σταθμούς ε, με ασφαλή τρόπο, περισσότερο από ό,τι ισχύει σήμερα. Αρχικά λοιπόν είχαμε πει ότι η ικανότητα θα μπορούσε να διπλασιαστεί ενώ θα διατηρείται η ασφάλεια του συστήματος. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο μας έχει απασχολήσει. Υπήρχε πρόταση της ε, ε, του φορέα μας, του οργανισμού μας, η Επιτροπή της περιέλαβε, υπήρχε διαπραγμάτευση στο Κοινοβούλιο και τώρα έχουμε το στόχο του 70%. Υπάρχουν λοιπόν ήδη ωφέλη προς τους ε, καταναλωτές. Βέβαια και πάλι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Θεωρούμε ότι αν ολοκληρώσουμε την αγορά της, την, την ολοκλήρωση της αγοράς ως διαδικασία, θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμα και ωφέλη 10 δις ευρώ κάθε χρόνο προς τους καταναλωτές στο φυσικό αέριο. Και πάλι βλέπουμε σημαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά το, τη συγκέντρωση κόστους ε, για την αγορά. Εδώ στους δύο χάρτες έχετε μια σύγκριση της κατάστασης το 2012 με το 2017. Σε κίτρινο βλέπετε την περιοχή όπου το συλλογικό κόστος ε, είναι πιο υψηλό και σε γαλάζιο λίγο λιγότερο. Βλέπετε ότι αυξάνεται η κίτρινη περιοχή, υπάρχει μεγαλύτερη ολοκλήρωση της αγοράς, επομένως οι καταναλωτές ε, εποφελούνται ε, αρκετά ανταγωνιστικού κόστους ε, απόκτησης. Μπορούμε λοιπόν, προσπαθούμε να προωθήσουμε την ολοκλήρωση της αγοράς και ότι αυτό αποδίδει. Δεν είναι πιο οικονομικό το φυσικό αέριο όταν είναι κοντά στην πηγή. Είναι φτηνότερο όταν είναι κοντά σε μια ανταγωνιστική αγορά. Και αυτό είναι σημαντικό. Θα ήθελα τώρα να επανέλθω ε, στον Acer. Αναφέρθηκα σε αρκετές ε, αποφάσεις ε, που έχουμε λάβει. Από κάτω προς τα πάνω λοιπόν, όταν οι εθνικές αριθμιστικές αρχές δεν ε, καταφέρουν να αποφανθούν ή όταν από κοινού αποφασίζουν να αφήσουν την απόφαση σε εμάς. Μέχρι τώρα έχουμε ε, λάβει πάνω από 15. Είχαμε στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς και αρχές της, αυτής είχαμε περίπου 20 και φυσικά σε εμά στέλνουν τις πιο σύνθετες και ακανθώδεις υποθέσεις, αλλιώς δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν και μόνοι τους. Υπάρχουν και άλλες αποφάσεις, αλλά δεν χρειάζεται να τα αναφέρω διεξοδικά. Τώρα, τελευταίος ε, τομέας αρμοδιοτήτων μας πριν περάσω στη δέσμη τη καθαρής ενέργεια. Λοιπόν, ο REMIT για την ενεργειακή αγορά, την ε, ακεραιότητα της αγοράς και τη διαφάνεια. Πρόκειται για κάτι άνευ προηγουμένου και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εποπτεία λοιπόν των συναλλαγών στην αγορά χονδρικής ε, της ηλεκτρικής ενέργειας. Της ενέργειας μάλλον ευρύτερα. Έχουμε λάβει λοιπόν ε, τα αρχεία όλων ε, των συναλλαγών εμπορίας ε, χονδρικής της ενέργειας. Έχουμε εντοπίσει κάποια μοτίβα ε, όπου θεωρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην αγορά. Έχουμε αναπτύξει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, μια πλατφόρμα που εξετάζει τα στοιχεία αυτά για να εντοπίσει κάποια, κάποια μη κανονικά στοιχεία τα οποία δεν είναι απαραίτητα προβληματικά, απλώς δεν είναι τα συνήθη. Και έχουμε λοιπόν μία ομάδα που εξετάζει ακριβώς αυτές τις περιπτώσεις για να δει κατά πόσο υπάρχουν υποψίες για κάτι χειρότερο. Λαμβάνουμε περίπου 3 εκατομμύρια αρχεία τέτοιων συναλλαγών ε, καθημερινώς, 70 με 80 λοιπόν εκατομμύρια κάθε μήνα, περίπου 10 με 12 χιλιάδες ε, τέτοια μη κανονικά ε, περιστατικά εξετάζουμε κάθε μήνα και περίπου 10% εξετάζει και να λέει η ομάδα μας στη Λουμπλιάνα, δεν μπορεί να κάνει παραπάνω. Το 90% λοιπόν αυτών των περιστατικών αυτή τη στιγμή δεν ελέγχεται. Και από τις 10-12.000 μάλλον από τα 1.000-1.200 τέτοια περιστατικά που ελέγχουμε, το 60-80% λέμε ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα και έτσι ε, μεταφέρονται προς την Εθνική Αρχή προς περαιτέρω διερεύνηση. Και εδώ έχετε ορισμένες ε, υποθέσεις που έχουν διερευνήσει οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές. Ε, αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι το βίντεο που είχαμε πέρυσι. Τώρα είναι σε μια διαδικασία έφεσης. Η Γαλλική Ρυθμιστική Αρχή λοιπόν είχε επιληφθεί ε, και είχε επιβάλει πρόστιμο 5 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα περνάω στη δέσμη για την καθαρή ενέργεια. Φαντάζομαι ξέρετε τα καθήκοντα που έχει αναλάβει ο Acer σε αυτό τον τομέα γιατί εσείς τα αποφασίσατε. Έχει λοιπόν ε, αρμοδιότητες για αρκετά κρίσιμη σημασία στέματα στην αγορά ενέργειας, επάρκεια πόρων, ετοιμότητα σε σχέση με κινδύνους, διασυνοριακή συμμετοχή, θετική έκπληξη μας προκάλεσαν αυτές οι αρμοδιότητες που μας εχωρίσατε και ελπίζουμε να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη θητεία. Έχουμε και επιπρόσθετες εποπτικές αρμοδιότητες για μία σειρά ε, ευρωπαϊκών ε, οντοτήτων, ένσω, περιφερειακά κέντρα συντονισμού και το καθεξής. Βασική πρόκληση είναι το γεγονός ότι πολλές από τις επιπρόσθετες αρμοδιότητες ενέχουν και προθεσμία που λύγει μέσα στους επόμενους μήνες. Μέχρι τώρα για φέτος έχουμε δοθεί μόλις 8 επιπρόσθετους ε, υπαλλήλους ενώ αρχικά είχαμε πρόταση για 28. Αυτό ήταν για μια ανάντη διαδικασία που περιλάμβανε και κριτήρια αναφορά benchmarking. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε, αλλά πραγματικά είναι πολύ δύσκολο γιατί απαιτεί πολλούς πόρους, ενώ ταυτόχρονα έχουμε και τις υπόλοιπες αρμοδιότητές μας. Λοιπόν, πόροι, πόροι, πόροι. Πρόσφατα μου ζητήθηκε να συντάξω ένα σύντομο άρθρο για την εμπειρία του οργανισμού και μου είπαν να εντοπίσω τρεις μεγάλες προκλήσεις. Ε, οι προκλήσεις αυτές είναι οι πόροι. Πόροι και πάλι πόροι. Γιατί από τότε που ετέθησε ισχύ το REMIT, ε, εμάς μας έχουν επιλήξει αυτοί οι ανεπαρκείς ε, πόροι. Και εδώ βλέπετε την διαφορά μεταξύ αυτών που έχουμε ζητήσει και αυτών που μας έχουν δοθεί. Μα λείπει περίπου το 1 τρίτο του απαιτούμενου προσωπικού. Δεν υπάρχουν προ το παρόν προοπτικέ. για το 2020, τουλάχιστον πριν την παρέμβαση του Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με την πρόταση τη Κομισιόν, λοιπόν, και πάλι θα μα λείπουν περίπου 40 άτομα. Μας απογοήτευσε το γεγονός ότι ότι δεν άνοιξε πάλι η πραγματεύση για το οικονομικό σκέλος, γιατί μας δόθηκαν ε, επιπλέον αρμοδιότητες και μάλιστα προτάθηκε εμείς να συνδράμουμε τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές σε ό,τι αφορά το REMIT. Από περιέργεια λοιπόν ζητήσαμε τις εθνικές αρχές τι θέλουν, σε τι θέλουν να τις βοηθήσουμε. Μας έδωσαν φυσικά ένα μακροσκελή ε, κατάλογο και όταν ε, ζητήσαμε επιπρόσθετους ε, πόρους μας έδωσαν μόλις 20, το οποίο δεν είναι λογικό. Λοιπόν, συμπερασματικά, μας τιμά ιδιαίτερα το γεγονό ότι μας έχετε χωρίσει νέες αρμοδιότητες, ιδίω σε πολύ κρίσιμους ε, τομείς με το πακέτο για την καθαρή ενέργεια. Όμως, αν δεν αλλάξει κάτι, εμείς δεν θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε. και για το REMIT είναι κάτι που μας δυσκολεύει γιατί πάλι βασίζεται στην αυτόματη διαλογή και εξέταση που βασίζεται σε μια πλατφόρμα που πάντα θα πρέπει να υποστηρίζεται. Από το 2016 έχουμε τριπλασιάσει τον αριθμό των ε, συναλλαγών που εξετάζουμε, αλλά και πάλι δεν έχουν αλλάξει οι πόροι μας. Βάσει της δική μας εκτίμηση και τη πρόταση τη Επιτροπή, το χάσμα μεταξύ των δύο λοιπόν είναι 4 εκατομμύρια, που δεν είναι τεράστιο ποσό στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για εμά θα κάνει όλη διαφορά. Τέλο, για την περίοδο 2021-2027. Η πρόταση Επιτροπή είναι 91 εκατομμύρια για την επταετία, δηλαδή 13 ε, έτο. Αυτό είναι κάτω και από αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για του χρόνου. Υπάρχει λοιπόν ε, σημαντική ανησυχία για την επιβίωση του οργανισμού μας μετά από το 2020. Πράγματι, υπάρχει διαδικασία και δυνατότητα επιβολής τελών για συγκεκριμένες λειτουργίες. Ελπίζω αυτό ε, να αρχίσει να λειτουργεί από το 2021. Φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι το κόλπο που θα ε, μας βοηθήσει να επιβιώσουμε και ελπίζω από κοινού με την Επιτροπή ε, να καταφέρουμε να διαμορφώσουμε αυτό το σύστημα Είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Διευθύντα. Πλήρης και πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση που μας δίνει μια εικόνα και της δουλειά σας και των προκλήσεων που έχετε μπροστά σας στην διεξαγωγή των δραστηριοτήτων σας. Μίλησαμε νωρίτερα για το θέμα του προπολογισμού και τα μέλη της Επιτροπής Εγγένεια να γνωρίζουν την ανάγκη να έχουν όλες οι υπηρεσίες ένα σωστό προπολογισμό και η δική σας ιδιαίτερα. Αυτό θα το αντικατοπτρίσει νομίζω και η γνωμοδότηση της Επιτροπής μας για τον προπολογισμό ότι δηλαδή χρειάζεται να έχετε έναν ουσιαστικό προπολογισμό. Συνάδελφοι, ποιος θέλει το λόγο. Καρβάλιο. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω καταρχά τον κύριο Ποτόσνικ για την παρουσίασή του. Πολύ καλή παρουσίαση. Η δουλειά της υπηρεσίας σας είναι εξαιρετικά σημαντική για το πακέτο ενέργειας. Οι ευθύνες της Επιτροπής σας αυξάνονται συνεχώς ιδίως τώρα με το νομοθετικό πακέτο για την καθαρή ενέργεια έχετε μεγάλη αύξηση των ευθυνών της υπηρεσίας σας. Όπως μας δείξετε, δεν έχετε επαρκείς πόρους και δημοσιονομικούς και σε ανθρώπινο δυναμικό και η κατάσταση δεν θα αλλάξει. Θα επιδεινωθεί μάλλον εν ώψη της επόμενης χρηματοδοτικής περίοδου 2021-2027. Η πρώτη μου ερώτηση λοιπόν είναι εσείς ως μάνατζερ, ως διευθυντής με εμπειρία τι πλάνα έχετε αν τα πράγματα δεν αλλάξουν. Δεύτερον, τεχνικό ερώτημα. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες για την παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς να τονίσω μια άλλη ευθύνη της υπηρεσίας που δεν σχολιάζεται πολύ. Την κατάσταση της ανάπτυξης των υποδομών. Πρόσφατα δημοσιεύσατε μια έκθεση με την κατάσταση των διαφόρων σχέσεων, των διασυνδέσεων, των σχεδίων κοινού, κοινού ενδιαφέροντος και διαπιστώσατε κάποιες καθυστερήσεις. Οι διασυνδέσεις είναι πολύ σημαντικές διότι μόνο με διασυνδέσεις ε, ολοκληρωμένες μπορεί να έχετε την πλήρως ε, ενοποιημένη αγορά προς όφελος των καταναλωτών και με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη. Ποιες είναι οι δυσκολίες, οι κύριες δυσκολίες. Να σας δώσω την περίπτωση της διασύνδεσης μεταξύ Ιβηρικής και Γαλλίας. Ισπανίας, Πορτογαλίας και Γαλλίας δηλαδή. το εγχείρημα αυτό τρενάρει εδώ και πολλά χρόνια και πάντα υπάρχουν δυσκολίες. Γιατί να υπάρχουν δυσκολίες σε κάτι που θεωρείται και τόσο εύλογο και τόσο σημαντικό για την εσωτερική αγορά για την ενέργεια στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Νίμπλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Πουτόσνικ για όλα αυτά που μας είπε. Ε, αφενός ε, μας παρουσιάσατε τον οργανισμό, τον Acer και μας δείξατε επίσης ε, το πώς θα προσαρμοστεί η Acer ως οργανισμό σε αυτό το νέο πακέτο Clean Energy, καθαρή ενέργεια. Και το είπατε πολύ σημαντικά ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τους, ε, την οικονομική στενοπό. Ε, μας τα επαναλάβατε όλα αυτά. Δύο ερωτήσεις έχω να σας κάνω. Η μία ερώτηση είναι η εξής. Νέες ε, προϋποθέσεις από το πακέτο καθαρής ενέργειας. Εμένα με ενδιαφέρει αυτός ο φορέας ο οποίος ε, ασχολείται με την διανομή και το δίκτυο διανομής αυτούς τους υποστηρίζετε ως φορέας. Και η δεύτερη ερώτησή μου αφορά την υποδομή, δαπάνες για την υποδομή. Η συνάλφος κυρία Καβάλιο ήδη το έθιξε το θέμα. Ίσως μπορείτε να είστε λίγο πιο συγκεκριμένος και όσον αφορά τις εργασίες σας. Ε, είχαμε πάρα πολλές ερωτήσεις σχετικά με την κατασκευή αγωγών και θέλω να ρωτήσω, ε, εσείς συμμετέχετε, νομίζω τον Απρίλη λάβατε μία απόφαση και όταν λαμβάνετε αυτές τις ε, αποφάσεις, τι κριτήρια εφαρμόζετε, αποδοτικότητα, εξοικονόμηση πόρων, ίσως μπορείτε να μας ε, βοηθήσετε να καταλάβουμε και εμείς πώς ακριβώς λαμβάνει ο οργανισμός σας αποφάσεις αυτής της εμβέλειας. Νομίζω αυτό θα μας βοηθούσε πάρα πολύ για να αξιολογήσουμε την εργασία σας. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ για την παρουσίασή σας κύριε Διευθυντά. Είδαμε πολλά θετικά στοιχεία από την υπηρεσία σας. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν εδώ ε, επιφυλάξει στην Επιτροπή. Αλλά είδα και πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζετε. Έλλειψη προσωπικού και επαρκούς χρηματοδότησης. Ελπίζω να πετύχουμε να αλλάξουμε τον πρώτο υπολογισμό και να βελτιώσουμε την χρηματοδότησή σας. Αλλά θα βρείτε προσωπικό έγκαιρα. Δεύτερη ερώτηση. Τα τέλη. Από ό,τι φαίνεται, δεν θα λυθεί η αύξηση των τελών μέσω και βράχη και μέσο πρόθεσμα. Η αύξηση των τελών, του κόστους χρήσης κάποιων υπηρεσιών θα καλύψει τα προβλήματα του προπολογισμού σα. τέλο πάντων, πρόθεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, η κυρία Φων Κράμον Ταομπαντέλη. Ε, να συνεχίσω εκεί που σταμάτησε η κυρία Νίπλερ. Εμένα με ενδιαφέρουν τρία θέματα. Το ένα είναι ότι μεταξύ άλλων αναφέρατε ότι με την αυξανόμενη διασύνδεση και με την επέκταση ε, των υποδομών η ε, τιμή του αερίου ανακάτοικο θα μειωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πολύ καλό, όμως εξακολουθούν να απομένουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Εμένα λοιπόν με ενδιαφέρει αφενός ε, η επέκταση των υποδομών, πώς προχωράει αυτό και οι συμβάσεις ε, που βρίσκονται πίσω από αυτή, την επέκταση. North Stream 2, ποιες είναι εκεί οι τιμές και με ενδιαφέρει επίσης ε, το ότι εφόσον πρόκειται για διμερείς ε, συμβάσεις, κατά πόσον αυτές έχουν προσαρμοστεί στην αγορά ενέργειας στην Ευρώπη. Και με ενδιαφέρει επίσης ε, την απόφαση του Διεθνικού Δικαστηρίου της Στοχόλμης από πέρυσι, ε, που καταδίκασε τη Ρωσία στην αντιπαράθεση με την Ναύτογκας όμως η Ρωσία αδιαφορεί. Ε, και εξακολουθεί να εκβιάζει την Ουκρανία με τέτοιο τρόπο που δεν μπορεί να μας εξυπηρετεί εμάς τους Ευρωπαίους. Με ενδιαφέρει ο δικός σας οργανισμός εμπλέκεται σε όλα αυτά ε, και πώς αξιολογείτε την έκβαση της υπόθεσης. Γιατί ξέρετε για την Ουκρανία υπάρχει μια στενοπός ενέργειας 7 κυβικά δισεκατομμύρια κυβικά και με το reverse flow δεν μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει στο να λυθεί το πρόβλημα. Ε, και υπάρχει κάποιο μοντέλο για κάποια άλλη λύση που προτείνεται. Έχετε ένα πρότυπο, ένα μοντέλο ή πρόκειται για ε, τυχαίες alerts, τυχαίες προειδοποιήσεις οι οποίες αποδεικνύεται ότι είναι και ανώδυνες. Okay, thank you. Someone else? Άλλος παρακαλώ. Ο κ. Ποτάσνικ. Well, thank you very much for very interesting questions and I was hoping for to be able to go back to some of the Um, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για αυτά τα θέματα που ε, θίξατε. Λοιπόν, θα τα πιάσω με τη σειρά. Επέκταση των ε, υποδομών. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειά μας αφορά την επέκταση των υποδομών. Υπάρχουν γενικές δραστηριότητες. Ο φορέας ε, γνωμοδοτεί ε, για ένα ε, δεκαετές πρόγραμμα το οποίο προετοιμάζει ένας φορέας για τη μετάδοση της ενέργειας. Επίσης, ε, γνωμοδοτούμε για θέματα κοινού συμφέροντος έτσι ώστε να έχουμε ε, ξεκάθαρα κριτήρια και να έχουμε και μία ε, ανάλυση κόστους ωφέλους. Άρα δηλαδή γνωμοδοτούμε για το κατά πόσον χρησιμοποιείται σε διάφορες περιοχές η ίδια μέθοδος. Αυτά καταρχήν ενίδιο, ε, μάλλον όσον αφορά τις γενικές μας αρμοδιότητες. Μετά ε, υπάρχει και μια γνωμοδότηση καταρχήν για τη Λιθουανία ε, και για ένα άλλο δίκτυο, LIPHOL, να καταναμηθεί το κόστος στις ε, διάφορες χώρες όταν δεν μπορούν να συμφωνήσουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Αυτά είναι λοιπόν τα, αυτά που κάνουμε κάθε χρόνο, οι γνωμοδοτήσεις. Πιο πρόσφατα ασχοληθήκαμε και νομίζω αναφερθήκατε σε αυτό σε μία απόφαση πολίτη για την διασύνδεση Ουγγαρίας-Αυστρίας. Εκεί λοιπόν είχαμε μια ελαφρά διαφωνία και πρέπει να το ξεκαθαρίσω γιατί υπήρξε μεγάλη σύγχυση και μέσα από τη διαδικασία έφεσης ε, που τρέχει τώρα στο ε, φετίο. Ε, το θέμα είναι ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει το αν είναι οικονομικά βιώσιμο όλο αυτό το σχέδιο, αλλά είναι δύο παράμετροι που πρέπει να εφαρμόζονται αν θα πρέπει να κατασκευαστεί ή όχι και δεύτερον υπό ποιε προποθέσει. Αυτές που ορίζει ο κανονισμός... πρέπει να υπάρχει ένα, μια δοκιμή στην αγορά και αν η αγορά ενδιαφέρεται να υπάρχουν οι υποδομές. Η διαφωνία που μας ε, επισημάνθηκε αφορά τις ε, παραμέτρους σχετικά με αυτή την δοκιμή στην αγορά. Οι δύο πλευρές ε, έχουν τελείως διαφορετική άποψη ως προς τις παραμέτρους που πρέπει να εφαρμοστούν. Τα υπόλοιπα καλύπτονται από τον κανονισμό. Ήθελα να το ξεκαθαρίσω αυτό. Τώρα, όσον αφορά το κατά πόσον τα τρέχοντα συστήματα είναι αποτελεσματικά ή όχι. Κοιτάξτε, εμείς ε, τοποθετούμε, τοποθετούμε τα για τα προγράμματα κοινού συμφέροντος κατά μέσο όρο 150, ε, με 50% των στα προγράμματα παρουσιάζεται καθυστέρηση. Υπήρξε κάποια πρόοδο τα τελευταία χρόνια, αλλά ακόμα υπάρχουν καθυστερήσεις. Ε, τα περισσότερα προγράμματα καθυστερούν στην αδειοδότηση. Ε, προσπαθούμε λοιπόν με τον νέο κανονισμό να εξορθολογήσουμε την όλη διαδικασία. Όλη η διαδικασία της αντιοδότησης δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 3,5 χρόνια και όλα αυτά αρχίζουν να αποδίδουν ε, αλλά ακόμα βέβαια δεν βλέπουμε απόλυτο εξορθολογισμό. Ε, τουλάχιστον δεν φαίνεται στα δεδομένα που μας αναφέρονται. Δεν βλέπουμε να υπάρχει σημαντική αλλαγή όσον αφορά την ανάπτυξη αυτών των προγραμμάτων. Κατά το υπόλοιπο μισή, εκεί προχωράμε κανονικά και αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Επίσης έχουμε την εντύπωση ότι τουλάχιστον αυτά τα ε, προγράμματα κοινού συμφέροντος σε αυτά ε, ορισμένα εξ αυτών είναι συμπληρωματικά αλλά είναι υποκατάστατα ως εκ τούτου ένα, ε, ένα πρόγραμμα που δεν προχωράει έγκαιρα αυτό πρέπει να το περιμένουμε και ελπίζουμε στον επόμενο γύρο που θα ακολουθήσει αργότερα. Ο φορέας που λαμβάνει τις αποφάσεις θα χρησιμοποιήσει την έκθεσή μας για να δει ε, σε ποια προγράμματα δεν σημειώνεται πρόοδος και θα το σκεφτούν ε, δύο φορές πριν ξαναπροτείνουν τέτοια προγράμματα ως προγράμματα κοινού συμφέροντος. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες μας ε, έναντι των χειριστών μετάδοσης, Αυτά ρυθμίζονται σε εθνικό επίπεδο από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Εκεί που υπήρχε κενό ε, και αυτό καλύφθηκε εν από το πακέτο ε, καθαρής ενέργειας, εδώ μιλάμε για τους ε, διανομής και τις αρμοδιότητές τους. Τώρα λοιπόν πράγματι η, ανάμεσα στις ε, εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τις ρυθμιστικές, τις ελεγκτικές αρχές υπάρχει μια συνεργασία, ε, θα έπρεπε να υπάρχει μια διαδικασία σαν αυτή που υφίσταται σε εθνικό επίπεδο, όπου η Εθνική ε, Ρυθμιστική Αρχή έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις και να τις κοινοποιεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, το πακέτο καθαρής ενέργειας. Ε, ε, εκεί είναι λίγο πιο περίπλοκο, αλλά είναι καλό το ότι σε τελική ανάλυση η απόφαση ανακοινώνεται στον φορέα διανομής. Για το προσωπικό, κατά πόσον αν υπάρχουν οι μπορούμε να βρούμε το απαραίτητο προσωπικό και αν θα βοηθήσουν τα τέλη. Κοιτάξτε, Είμαστε αρκετά τυχεροί. Έχουμε βρει καλό προσωπικό που δουλεύει για μας και για όσους ενδιαφέρονται για τον κανονισμό της ενέργειας. Η ενέργεια είναι σημαντική όταν πρόκειται για τον έλεγχο της αγοράς, γιατί από εκεί βλέπει κανείς το σύνολο της Ευρώπης. Έχουμε λοιπόν πολλούς ε, παθιασμένους ε, συναδέλφους. Αυτή τη στιγμή Έχουμε ελλείψεις βέβαια και αν μας δώσετε τη δυνατότητα να προσλάβουμε περισσότερο προσωπικό θα το πράξουμε. Ξέρετε βέβαια καλύτερα από μένα ότι περισσότερα χρήματα ε, δεν σημαίνει απαραίτητα και περισσότερο προσωπικό. Τα τέλη είμαι αισιόδοξο. Ε, με έχουν ρωτήσει ε, ποιο είναι το πρόγραμμά μου. Κοιτάξτε, το πρόγραμμά μας αυτή τη στιγμή είναι να επιβάλλουμε τέλη, γιατί δεν έχουμε άλλη δυνατότητα να πείσουμε τις δημοσιονομικές αρχές να αντιστρέψουν την τάση. Γιατί η άλλη εναλλακτική λύση είναι να παρετηθούμε ή ε, να μας δώσουν τα τέλη. Δουλεύουμε λοιπόν πάνω σε αυτό, στα τέλη. Ελπίζουμε τα τέλη να ισχύσουν από την επόμενη χρονιά, το πολύ πολύ το 2021 τα τέλη θα εξετάσουν και θα αντιμετωπίσουν ε, κάποια ε, προγράμματα όπου χρειαζόμαστε χρηματοδότηση. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα περισσότερο προσωπικό και μετά πρέπει να ξεκινήσει το σχέδιο ανάκαμψης. Ε, στο πακέτο καθαρής ενέργειας υπάρχει μία πρόβλεψη ότι μετά από ένα χρόνο η Κομισιόν θα εξετάσει τις ανάγκες σε χρήματα. Ε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Η, όλη οι επιπρόσθετοι πόροι θα προκύψουν το 22-23. Όπως σας είπα όμως το κλειδί είναι η επόμενη χρονιά. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ελπίζουμε τουλάχιστον για του χρόνου να έχουμε περισσότερο προσωπικό και πόρους που θα προέρχονται από τον ενωσιακό προϋπολογισμό. Τώρα, ε, μακροπρόθεσμα, αν δεν αλλάξει το πολιτεύσιμο δημοσιονομικό πλαίσιο, είμαστε αναγκασμένοι να εξαρτώμεθα από τα τέλη. Και πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά τους φορείς της αγοράς, οι φορείς της αγοράς το δέχονται. Όταν ξεκινήσαμε αυτές τις ε, διαδικασίες REMIT, ε, πολλοί ξεπλάγησαν παραδείγματο χάρη για τις αναφορές ε, στην ΕΣΜΑ ε, πρέπει να καταβάλλεται τέλος. Άρα δηλαδή οι ε, φορείς είναι προετοιμασμένοι. Το δικό μας το τέλος θα είναι πάρα πολύ μικρό, ποσοστιαία, δεν θα τους επηρεάσει. Δεν μιλάμε για μεγάλη συνεισφορά, μεγάλο υψηλό τέλος. Νομίζω ότι θα με συγχωρήσετε αν δεν μπω τόσο πολύ στις σχέσεις με τρίτες χώρες. Ο φορέας μας ε, δεν έχει εντολή ε, για να δραστηριοποιείται πέρα από τα σύνορα. Έτσι, North Stream και Ουκρανία, αυτά τα θέματα ε, καλύτερα να τα απαντήσει η Κομισιόν. Αλλά βλέπετε ότι η Ουκρανία ε, τροφοδοτείται τώρα από τη Δύση, ίσως με ρωσικό αέριο, αλλά από τη Δύση. Κάτι που πριν από 10 χρόνια δεν ήταν δυνατόν. Και αυτή είναι η προσπάθεια του Ευρωπαίου νομοθέτη για όλες τις διασυνδέσεις στην Ευρώπη, αυτό να είναι δυνατόν γιατί αυτό ε, όχι μόνο βοηθάει στο να υπάρχει ασφάλεια εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στους γείτονές μας. Και αυτό είναι πάλι ένα χειροπιαστό όφελος για τους πολίτες μας και αυτούς των γειτονικών χωρών. Και όσον αφορά τέλος ε, της προειδοποίησης, τα alert, ε, σας είπα αυτή τη στιγμή μπορούμε να ελέγχουμε το 10% των ανομαλιών έχουμε ένα αυτόματο σύστημα και μάλιστα προσπαθούμε να ιεραρχήσουμε με βάση τη συχνότητα και τις ε, επιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, αν δείτε κάτι το οποίο δεν είναι πολύ μεγάλη σημασία, τότε ε, δεν το εξετάζουμε περαιτέρω, αλλά είναι κάτι που είναι επαναλαμβανόμενο ή που προκαλεί σημαντική ζημιά στην αγορά, τότε το ιεραρχούμε και όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή ε, είμαστε σε θέση να αναλύουμε περίπου το 10% αυτών που μας αναφέρονται από τον έλεγχο ως ανομαλίες. Βέβαια, ε, μου λένε παραπονιέσαι ότι δεν έχετε χρήματα και παρόλα αυτά είστε αποτελεσματικοί. Ε, εμείς λέμε, το 10% αλλά μάλλον εξετάζουμε το 10% αλλά δεν λέμε ποιο είναι αυτό το 10%. Άρα οι φορείς ε, εμπλεκόμενοι δεν ξέρουν αν τους ελέγχουμε ή όχι. Με αυτό το πακέτο της καθαρής ενέργειας και με τις νέες αρμοδιότητες ε, θα είμαστε πιο ορατοί Υποτίθεται ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει μια έκθεση βέλτιστων πρακτικών για τους στόχους μετάδοσης ε, ηλεκτρικής ενέργειας. Με τους πόρους που έχουμε είναι πολύ δύσκολο να καταθέσουμε μια έκθεση βέλτιστων πρακτικών. Αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι συγκεντρώνουμε πληροφορίες από τα κράτη-μέλη ε, και καταθέτουμε μια έκθεση αυτό ίσως να απογοητεύει εκείνους που μας έχουν δώσει την εντολή. Ίσως ναι, ε, μέχρι τώρα δεν ήμασταν τόσο ορατοί, αλλά προφανώς ήδη τώρα ε, δεν μπορούμε να είμαστε τόσο αποτελεσματικοί όσο θα θέλαμε. Γι' αυτό είμαι ευγνώμων για τις προσπάθειές σας. Η Πρόεδρος είπε ότι θα στηρίξει ε, τον οργανισμό μας και αυτό για μας ε, είναι μια πολύ μεγάλη παρηγοριά γιατί πολλές φορές βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Ευχαριστούμε. Πραγματικά οι απαντήσεις ήταν όλες ε, πολύ ενδιαφέρουσες. Είδαμε από μέσα όλα τα ζητήματα ενέργεια, αγοράς ενέργειας στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον και καινούργια πράγματα για πολλούς από εμάς. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και όπως σας είπα προσπαθούμε να υποστηρίξουμε την υπηρεσία σας και τις καινοτόμες πρακτικές σας για να λύνει τα προβλήματα χωρίς έναν ουσιαστικό προϋπολογισμό. Ελπίζουμε ότι αυτό θα λήξει και θα μπορέσουμε να σας δώσουμε περισσότερα κονδύλια για την υπηρεσία. Περιμένουμε την έκθεση βέλτιση των πρακτικών του χρόνου. Ευχαριστούμε. Um, uh, uh, uh, Ο κ. Ποτόσνικ ε, μας ενημερώνει ότι η παρουσίαση είναι διαθέσιμη, μπορεί να την πάρετε έξω, στην είσοδο δηλαδή. Uh, Επόμενο θέμα. Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή για την ΕΝΙΖΑ. Κυβερνοασφάλεια και ΕΝΙΖΑ. Καλέσαμε την κυρία Δέσποινα Σπανού, Διευθύντρια, Γενική Διευθύντρια στη DG Connect. Καλώς ήρθατε. Χθες συνάντησα τον ε, προτινόμενο εκτελεστικό διευθυντή της ΕΝΙΣΤΑ, τον κύριο Λεπάσαρ. Συμφωνήσαμε να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων μαζί του για να οργανώσουμε την ακρόαση για τη θέση του το Σεπτέμβριο και με την ευκαιρία αυτή θεώρησε ότι ήταν σκόπο να έχουμε μια συζήτηση και με την DG Connect για να συζητήσουμε εκτενέστερα το περιβάλλον κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη και το ρόλο της ΕΝΙΖΑ στο πλαίσιο αυτό. Η κυρία Σπανού λοιπόν έχει το λόγο για να παρουσιάσει αν θέλετε τα δεδομένα και να κάνουμε έναν ουσιαστικό διάλογο. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ευχαριστούμε που, μας καλέσατε, που με καλέσατε στην συνάντηση αυτή. Να καλωσορίσω και τα καινούργια μέλη, να καλωσορίσω και αυτούς που επανέρχονται. Ο τομέας της κυβερνοασφάλειας τα τελευταία χρόνια ήταν ε, σημείο έμφασης κομισιών. Είχαμε και έναν κανονισμό για την κυβερνοασφάλεια, ένα θετικό κείμενο για την κυβερνοασφάλεια. Ε, παίξει καθοριστικό ρόλο στη, στο κείμενο αυτό. Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο και τέθηκε σε ισχύ το νομικό αυτό κείμενο 27 Ιουνίου. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες λοιπόν μπήκαμε σε, ένα νέο, σε μια νέα εποχή ασφάλειας. Το κείμενο πρώτον αναθεωρεί την εντολή της ΕΝΙΖΑ και εισάγει το πρώτο ιστορικά πλαίσιο πιστοποίησης. Να κάνω μια σύντομη ενημέρωση του τι κάνει η Ενίζα και από πότε και τι αλλαγές έγιναν με το πρόσφατο αυτό νομοθετικό κείμενο του Cyber Security Act για να έχετε μια εικόνα. Μια και θα συνεργαστούμε τα επόμενα χρόνια. Η ιστορία της Ενίζα ξεκινά το 2004 με τον κανονισμό θέσπισής της που δημιούργησε μια τυπική αποκεντρωμένη υπηρεσία που θα υποστήριζε τα κράτη-μέλη σε ζητήματα ασφάλειας των πληροφοριών και των πληροφοριακών συστημάτων. Αυτό ήταν η πρώτη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει μια ανεξάρτητη υπηρεσία με, χωρισ... με ιδιαίτερη διαχείριση από τα κράτη-μέλη με τη συνεργασία και τις Επιτροπής που θα υποστήριζε τις προσπάθειες να επεκταθεί η γνώση που έχουμε στην Ευρώπη για την κυβέρνηση ασφάλεια ένας τομέας όπου η γνώση είναι δυναμική γιατί εξελίσσεται κάθε μέρα και την βελτίωση των ικανοτήτων των κρατών μελών. Αυτή η πρώτη εντολή του ΕΝΙΖΑ είχε ένα ειδικό χαρακτηριστικό που δεν το βρίσκεται σε άλλες υπηρεσίες. Δεν ήταν μόνιμη υπηρεσία. Είχε προθεσμία λήξης και επεκτάθηκε η λειτουργία της δύο φορές, το 2008 και το 2000, το 2011 ως και το 2013 ο κανονισμός επεξέτεινε την, επε, ε, την εντολή της ε, ε, υπηρεσίας για άλλα 7 χρόνια ζητώντας να κάνει μια πλήρη αξιολόγηση της δουλειάς της πριν λήξει αυτή η περίοδος και να προτείνει για το κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει μόνιμη ή όχι. Για το λόγο αυτό το 2017 κάναμε μια πλήρη αξιολόγηση με υποστήριξη εξωτερικής ανεξάρτητης μελέτης όλα τα στοιχεία της υπηρεσίας και προτείναμε στο νομοθετικό αυτό κείμενο να γίνει μόνιμη η εντολή για την ΕΝΙΖΑ. Τώρα, Ποια ήταν τα αρχικά της κατηθήκοντα. Η αποστολή δεν άλλαξε. Είναι να συμβάλλει σε υψηλό επίπεδο ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια, ο στόχος ήταν μια ευέλικτη υπηρεσία. Είναι μικρή, έχει 80 άτομα προσωπικό πλήρους απασχόλησης και συνεργάζεται στενά με τους ειδικού των κρατών μελών αλλά και με τον ε, ιδιωτικό τομέα, με τον κλάδο που έχει και πολλή γνώση αλλά και υφίσταται και πολλές επιπτώσεις από τις παραβιάσεις ε, ασφάλειας ε, στην Ένωση. Στην Ελλάδα είναι εγκατεστημένο, τίποτα δεν έχει αλλάξει αυτά τα χρόνια. Η τομή δουλειά τη ΕΝΙΖΑ τα τελευταία χρόνια ήταν να, δώσει, να δώσει τα κράτη-μέλη και στου ευρωπαϊκού θεσμού υψηλή εμπειρία στον τομέα τη ασφάλεια, έναν τομέα όπου υπήρχε ένα πρόβλημα γνώσεων, δεξιοτήτων και κατανόηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μελέτε, με συνεργασία με του διάφορου εμπλεκόμενου φορεί, να βοηθήσει τα κράτη-μέλη και τις, ε, τα, θεσμικά όργανα στην ενίσχυση των, αντι, των πολιτικών κατά τη ε, κυβερνο, κυβερνοπαρέμβασης. Η οδηγία που τέθηκε σε ισχύ πέρσι δημιούργησε ένα ολόκληρο σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισης ε, της κυβερνοασφάλειας. Η Ενίζα παρέσχε συμβουλευτική, διότι εξέφεσε στα κράτη-μέλη το πώς θα λειτουργούσαν, αλλά πήρε και έναν ειδικό ρόλο, διότι η Ενίζα ήταν μέλος όχι μόνο του δικτύου αλλά και της ομάδας που προετοίμαζε τα κείμενα. Επίσης, η Ενίζα έχει αρμοδιότητα να βοηθήσει τα κρατημένα να αναπτύξουν τις δικές τους ικανότητες αντιμετώπισης της κυβερνοασφάλειας και έχει και συνεργασία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι για να ξέρουμε τι, γιατί είναι γνωστή η Ενίζα. Πρώτα, Cyber Europe, εξαμηνιαία άσκηση κυβερνοασφάλειας που γίνεται εδώ και κάποια χρόνια, το δημιούργησε η ΕΝΙΖΑ. Σε αυτήν μετέχουν όλοι οι πυρογνώμονες των κρατών μελών και λειτουργούν προστατεύοντας από επίθεση και δίνοντας και απαντώντας από κοινού. Αυτό επιτρέψει, επέτρεψε τα κρατημέλη να βρουν πού είναι οι τροτότητέ του, ενίσχυσαν να ενισχύσουν τι δυνατότητε του, αλλά κυρίω έφερε τα κράτη-μέλη σε ένα σενάριο πραγματική ζωή όπου υπάρχει μια ε, μαζική κυβερνοεπίθεση και το πώ μπορούν να συνεργαστούν τα κράτη-μέλη. Ούτω ή άλλω, οι περισσότερε κυβερνοεπιθέσει έχουν αντικτύπους και αλλού και να δουν τι δυνατότητε απάντηση. Η Ενίζα κάθε Οκτώβριο κάνει τον μήνα κυβερνοασφάλειας. Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου γίνεται μια καμπάνια ενημέρωσης που συντονίζει η ΕΝΙΖΑ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου γίνεται ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών, μεταξύ ιδιωτών, μεταξύ ερευνητικών Ινστιτούτων για όλα τα συστήματα όχι μόνο τον κλάδο και για τους πολίτες, για τους φοιτητές τους, ώστε να έχουν καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων της κυβερνοασφάλειας σε έναν ολοένα και πιο ψηφιοποιημένο κόσμο. Επίσης, η ΕΝΙΖΑ οργανώνει την πρόκληση, το Cyber Security Challenge όπως το λένε. Ένας διαγωνισμός μεταξύ νεαρών φοιτητών, μαθητών ανά την Ευρώπη που, για τα θέματα κυβερνοασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τη γνώση και την ενίσχυση των δυνατήτων, η ενίσχυση είναι γνωστή ανά τον κόσμο για το τοπίο απειλών, threat landscape που δημιουργεί. Ένα πληρέστατο κείμενο που παρέχει τις ε, απειλές και τους αναδυόμενους κινδύνους, ε, παρέχοντας πληροφορίες σε και στον κλάδο. Ταυτόχρονα από την υιοθέτηση του κανονισμού ΕΝΕΣ μετέχει στο δίκτυο ΣΥΣΕΤ, παρέχει την γραμματιακή υποστήριξη που είναι ένα, αυτό είναι ένα δίκτυο όλων των ομάδων άμεσης ανταπόκρισης σε περίπτωση κυβερνο, κυβερνοεπίθεσης. Έχει έναν ρόλο δηλαδή συντονιστή σε μια τέτοια κατάσταση. Όλα αυτά παραμένουν στον, στην έντολη της ΕΝΙΖΑ. Προστίθενται όμως και κάποια σημαντικά στοιχεία. Πρώτον, η εντολή γίνεται πολύ πιο στοχοθετημένη. Η αξιολόγηση έδειξε ότι η Ενίκη είναι μια μικρή υπηρεσία. Είναι πολύ λοιπόν σημαντικό να έχουμε λεπτομεριακή περιγραφή των καθηκόνων τη ώστε να τα ε, υλοποιεί. Επίσης ήταν σαφέ ότι η Ενίσα δεν μπορούσε να καλύψει με τους πόρου που είχε, άρα χάρη στο Cyber Security Act και την επιτροπή σας που μας, που μας υποστήριξε, έχουμε αύξηση του προσωπικού του ΕΝΙΖΑ. 84 άτομα είναι τώρα, 125 θα είναι τα επόμενα έτη, μέσα στα επόμενα 4 έτη. Και ο προπολογισμό θα διπλασιαστεί από 11 σε 23 εκατομμύρια την επόμενη τετραετία. Κάτι ακόμα πιο σημαντικό, ο κανονισμός παρέχει μία μόνιμη εντολή, δηλαδή γίνεται μόνιμη υπηρεσία χωρίς να ε, αλλάζοντας δηλαδή την προγενέστερη κατάσταση. Διακυβέρνηση, διοίκηση δηλαδή. Και εδώ η ΕΝΙΖΑ είναι λίγο διαφορετική από τις άλλες υπηρεσίες. Υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο 30 μελών. Τα 30 μέλη περιλαμβάνουν 28 εκπροσώπους από τα κράτη-μέλη, από τις κρατικές υπηρεσίες και 2 από την Επιτροπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το Management Board, έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο διότι εγκρίνει όλες τις αποφάσεις που σχετίζονται με την ε, υπηρεσία, τον προγραμματισμό που εγκρίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποστηρίζεται από ένα εκτελεστικό γραφείο, ένα μικρότερο όργανο που επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει την ευθύνη της ε, των εκτελεστικών δραστηριοτήτων της ε, ε, ΕΝΙΖΑ. Υπάρχει και ένα σύστημα εθνικών αξιωματικών συνδέσμων που λειτουργούν ως δίκτυο διαμόρφωσης πολιτικής για τη συζήτηση των βασικότερων ε, θεμάτων πολιτικής με, που, με, τα οποία ασχολείται η ε, ΕΝΙΖΑ. Μέχρι το προγενέστερο νόμο ήταν ένα ad hoc όργανο, τώρα μπορεί να γίνει μόνιμο. Έχουμε και τον εκτελεστικό διευθυντή που είναι ο επικεφαλής της ε, υπηρεσίας. Έχει μια συμβουλευτική επιτροπή που ήταν η μόνιμη επιτροπή εμπλεκομένων που με τον καινούριο Cyber Security Act παίρνει το όνομα Permanent Advisory Group, μόνιμη ε, συμβουλευτική ομάδα. Ορίζονται μετά από πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή από το Διοικητικό Συμβούλιο και του παρέχουν ad personam, ad personam συμβουλευτικές δραστηριότητες. Είναι άτομα δηλαδή με ειδικές γνώσεις που παρέχουν συμβουλές στον ίδιο τον εκτελεστικό διευθυντή. Δεν είναι ένα θεσμικό όργανο, είναι μια ομάδα εμπλεκομένων φορέων που λειτουργεί ad hoc. Και έχουμε και το προσωπικό του ΕΝΙΖΑ που αυτή τη στιγμή ε, ε, ε, είναι μοιρασμένο σε μια σειρά διοικητικών δομών. Ορισμός του εκτελεστικού διευθυντή. Αυτό ήταν και το ξεκίνημα της συζήτησης. Να σας εξηγήσω τι λέει το Cyber Security Act, ο νόμος ασφάλειας Δεν διαφέρει σε σχέση με τον προηγούμενο κανονισμό. Ο εκτελεστικός διευθυντής ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η, η, αρχή, η υπεύθυνη αρχή πρόσληψης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση πρόταση της Επιτροπής. Η Επιτροπή ε, πρέπει να επιλέξει μια shortlist, ένα ε, πρώτο κατάλογο για την εκλογή του διευθυντή χρειάζεται πλειοψηφία δύο τρίτων θητεία πενταετής το νομοθετικό κείμενο ε, ο νόμος για την κύβερνο ασφάλεια προβλέπει ότι ο εκτελεστικό διευθυντή πριν την ε, τοποθέτησή του πρέπει να κάνει μια δήλωση στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εσάς δηλαδή, και απαντά και στα κρατημέλη. Αυτή ήταν η διαδικασία της ακρόασης που ανέφερε νωρίτερα η πρόεδρος για το Σεπτέμβριο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο θα προχωρήσει επίσημα στον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή η θητεία του οποίου λήγει στις 15 Οκτωβρίου. Για να υπάρξει καλή συνέχεια της υπηρεσίας θα ήταν σκόπιμο μετά τις 15 Οκτωβρίου να έχουμε ήδη το νέο εκτελεστικό διευθυντή και η απόφαση λήφθηκε την περασμένη εβδομάδα γρήγορα γρήγορα. Μετά η Επιτροπή έχει υιοθετήσει το shortlist το Μάιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν αποφασίσει να επεκτείνει την θητεία του, του εκτελεστικού θητή μετά το τέλος της θητείας. Τώρα για το timing, να σας πω ότι έπρεπε να περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις ε, του νόμου κυβερνοασφάλειας πριν ξεκινήσει μια νέα διαδικασία, διότι μέσα στην, ε, στο νομοθετικό κείμενο υπήρχαν θέματα που έπρεπε να λυθούν γιατί αφορούσαν τον ορισμό του εκτελεστικού διευθυντή, θητεία κλπ. Άρα έπρεπε να κλείσει ο νόμος για να προχωρήσουμε στη νέα επιλογή του ε, εκτελεστικού διευθυντή. Από το Δεκέμβριο δηλαδή μέχρι το Μάιο προχωρήσαμε για την ε, ανακοίνωση της κλπ. Τώρα, τι, ποια είναι τα νέα καθήκοντα της ΕΝΙΖΑ μετά τις 27 Ιουνίου και τι θα πρέπει να υλοποιήσει ο νέος εκπαιδευτικός διευθυντής. Ανάπτυξη πολιτικής και εφαρμογή τους. Αυτό το έκανε εξ αρχή η ΕΝΙΖΑ από την δημιουργία της, αλλά έκτοτε έχουν υιοθετηθεί νέα νομοθετικά κείμενα που προσφέρουν πολλά καθήκοντα η εφαρμογή της, του κανονισμού για την ηλεκτρονική ταυτότητα, οδηγία ENS, ε, μια σειρά νέων στοιχείων δηλαδή. Υπάρχει ευθύνη για την εφαρμογή της οδηγίας για το ENIS, ε, σε στενή συνεργασία δηλαδή η ΕΝΙΣΑ συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη για τον ε, σχεδιασμό των προτύπων και πρέπει να παράσχει μια ετήσια έκθεση για την εφαρμογή, την κατάσταση εφαρμογής ε, του νομοθετικού πλαισίου για την κυβερνοασφάλεια. Ε, κάνει δηλαδή και επανεξέταση του πλαισίου, του νομοθετικού πλαισίου. Επίσης, ό,τι αφορά το capacity building, ε, η ΕΝΙΖΑ υποστηρίζει την ενίσχυση των ικανοτήτων των κρατών μελών και μετά το νέο νομοθετικό κείμενο έχει και την ευθύνη για την ανάπτυξη ενός συστήματος αντιμετώπισης ε, ε, διαπίστωσης των τοτήτων. μια νέα αρμοδιότητα που προέκυψε μετά από δικό σας έτοιμο όταν ζητήσατε να έχετε μια πολιτική ε, αποκάλυψη των τοτήτων ως πλαίσιο για την διαμόρφωση μιας κουλτούρας αμοιβαίας ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών. Επίσης κάνει και τις ευθύνες της αναθεώρησης των εθνικών και των κοινωνικών πολιτικών. Ακόμα πιο σημαντικό η νέα νομοθεσία ασφάλειας προσθέτει καθήκοντα στην έννοια ότι αφορά την επιχειρησιακή συνεργασία. Το άρθρο 7. Η ΕΝΙΣΑ όχι μόνο έχει λοιπόν την, τις παλιές ευθύνες, τη γραμματιακή υποστήριξη δηλαδή του συντονιστικού, τώρα έχει και την ευθύνη σε περίπτωση μαζικής μεγάλης κυβερνοεπίθεσης να ετοιμάσει μια έκθεση επίγνωσης και έκθεση κατάστασης και μπορεί τα κράτη-μέλη να ζητήσουν από την ΕΝΙΖΑ να παράσχει πραγματική υποστήριξη. Επιπλέον είναι υπεύθυνη να παράσχει μία μόνιμη τακτική έκθεση καταστάσεων και αντιμετώπιση των προβλημάτων να δημιουργεί, να λειτουργήσει δηλαδή ως ένα κεντρικό ε, σημείο αναφοράς πληροφοριών. Αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια. Κλείνω εδώ, Πρόεδρε. Παρέχει υποστήριξη σε ex τεχνική έρευνα. Αν γίνει δηλαδή σήμερα μια γενική ε, κυβερνοεπίθεση δεν έχουμε το πλαίσιο για να κάνουμε μια τεχνική μελέτη για το πώς έγινε. Η Ενίζα με το νέο νόμο μπορεί να το κάνει και θα πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσει τις ε, ικανότητες που έχει για να λειτουργήσει μέσω του, για, την, ε, λειτου, να λειτουργήσει το blueprint, δηλαδή έναν κώδικα του ποιος κάνει τι σε περίπτωση ε, κυβερνοεπίθεσης το blueprint λοιπόν πρέπει να αναπτύξει αυτές τη, με βάση το blueprint πρέπει να αναπτύξει μια σειρά ε, καθηκόντων και να εφαρμόσει το CETU που είναι η ομάδα ανταπόκρισης. Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές του, της νομοθεσίας για την κυβερνοασφάλιση είναι οι ευθύνε για το σύστημα πιστοποίηση που δημιουργήθηκε με το νόμο αυτό. Είναι το πρώτο πλαίσιο πιστοποίηση που υπάρχει στην ιστορία τη Ένωση. Για συνδεδεμένα προϊόντα και συστήματα δεν είχαμε μέχρι την, ε, το, νόμο για την κυβερνοασφάλεια νομοθετικό πλαίσιο. Δηλαδή για την ασφάλεια των προϊόντων ICT. Αυτό είναι ένα πλαίσιο εθελούσιο, καλύπτει τομείς αγοράς που θεωρείται ότι είναι αναγκαίο περισσότερο και στο κέντρο αυτής είναι η Νίζα διότι παρέχει τα προγράμματα που θα γίνουν με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και θα εφαρμοστούν ε, συνολικά στην Ευρώπη. Αυτό το πλαίσιο πιστοποίησης καλύπτεται από το σύστημα ε, επιτροπής συμβουλευτικής από πλευράς κρατών μελών και εμπλεκομένων φορέων που μαζί συμβουλεύουν την ΕΝΙΖΑ και η ΕΝΙΖΑ θα πρέπει να ξεκινήσει να κάνει την αξιολόγηση των προγραμμάτων με πρότυπα, με εμπλεκόμενους κλπ. Μιλάμε για πολλή δουλειά. Ε, ένα μεγάλο κομμάτι των πόρων της ΕΝΙΖΑ πήγε σε αυτό το σκοπό και ήδη έχει ξεκινήσει η επιστοποίηση της, από πλευράς ΕΝΙΖΑ σε κάποιους τομείς. Αυτό ίσως είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχει να κάνει τι αμέσω επόμενες μέρες θα έλεγα η Ενίσα. Εναρμόνιση και αυτό σχετίζεται με την πιστοποίηση και τόνισα νομίζω και το ρόλο της Ενίζα να δημιουργήσει ένα παρατηρητήριο αγοράς που εξετάζει τις ε, τάσεις στην ε, στην αγορά Αυτά για τα νέα καθήκοντα της Ενίζα Πρόεδρε, στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρουσίαση ιδιαίτερα επίκαιρη. Ήδη οι συνάδελφοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να πάρουν το λόγο. Η κυρία Νίμπλερ πρώτη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμη κυρία Σπανού. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα στην Επιτροπή μας ε, και θα ήθελα αυτής εξ αρχής ε, να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ε, θα μας δοθεί δυνατότητα να δούμε ε, τον νέο διευθυντή της ΕΝΙΑ, τον κύριο Πασάλντο, ε, είχα την εντύπωση ότι θα ερχόταν σήμερα, αλλά αφού θα αναλάβει τον Οκτώβρη, να έρθει το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε και η μετάβαση να είναι και χωρίς προβλήματα. Πρώτη παρατήρηση αφορά στη νέα επιτροπή. Νομίζω ότι το θέμα της κυβερνοασφάλειας είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και χαίρομαι πάρα πολύ, κυρία Σπανού, για το γεγονός ότι με την πράξη κυβερνοασφάλειας και με την ΕΝΙΖΑ ε, πλέον μπορούμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Κατά την προηγούμενη θητεία, ακριβώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε δώσει μεγάλη σημασία έτσι ώστε η ΕΝΙΖΑ να μην είναι μόνο μια γραμματεία για τα κράτη-μέλη ή για την Επιτροπή, αλλά και διακομματικά να μπορεί κανείς να απευθυνθεί στην Επιτροπή, η Επιτροπή να είναι ανεξάρτητη, να έχει τα δικά της καθήκοντα. Ε, μιλήσατε operational cooperation. Αυτό το θέμα για μας ήταν πολύ σημαντικό όπως επίσης και η συμπερίληψη της ΕΝΙΖΑ ε, σε προετοιμασίες για τυποποίηση ε, κυρίως ε, για το ε, Candidate Security Scheme. Αυτό είναι μία από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες της ΕΝΙΖΑ για τα επόμενα έτη. Και να ξέρετε, θα μας βρείτε στο πλευρό σας, θέλουμε να στηρίξουμε την ΕΝΙΖΑ. C, αυτό είναι το θέμα που απασχολεί όλα τα κράτη-μέλη και σε όλα τα κράτη. μελη Για το 5G, 5G έχουν ξεκινήσει οι διαγωνισμοί και από ό,τι θυμάμαι η Κομισιόν ε, έχει ε, τοποθετηθεί και αυτή για το δίκτυο 5G, 5G. Και ενώ εσείς, ερωτώ, εσείς τι κάνετε, συντονίζετε τα κράτη-μέλη για το δίκτυο 5G. Και επίσης ε, ε, το πρώτο σύστημα πιστοποίησης ε, για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί στο σύστημα 5G. Ε, τι ακριβώς έχετε να μας πείτε από αυτού. Και το δεύτερο ερώτημα είναι πολιτικής φύσεως. Θα ήθελα να μας πείτε τη γνώμη σας. Ψηφιακή κυριαρχία της Ευρώπης. Συζητιέται παντού. Και είναι πολύ σημαντικό το να δει κανείς ότι έξω ευρωπαϊκή φορείς αρχίζουν να κυριαρχούν στην ευρωπαϊκή αγορά και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ρωτώ, εσείς τι σκέπτεστε, η γενική σας διεύθυνση τι έχει κατά νου ε, σε σχέση με αυτό το θέμα των ευρωπαϊκών προμηθευτών. Ίσως μπορείτε να τοποθετηθείτε από αυτού. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Καλυμπράντη. Ευχαριστώ για την εξαιρετική παρουσίαση. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σας άκουσα. Και προσβλέπω και στη συζήτηση με τον κύριο Λεπασά, που σίγουρα θα ε, είναι πολύ μεγάλο ατού για την Ενίζα και εξαιρετικός ε, διευθυντής. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν τα όσα είπατε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ που παρουσιάσατε και δημοσιεύσατε το έγγραφο πολιτικής ε, που προαναφέρατε, που λέει και για την ψηφιακή ε, κυριαρχία. Ήθελα λοιπόν να σταθώ σε αυτό το ζήτημα, γιατί ξέρω ότι είναι ένα πολύ ακαθόδε ζήτημα στο διεθνές στερέωμα. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτό το προηγούμενο ερώτημα, σίγουρα θα το ε, απαντήσετε. Όμως ένα ευρύτερο ερώτημα τώρα για τη συνεργασία και μάλιστα τη διεθνή συνεργασία. Από την παρουσίασή σα, ε, είδα πως η ΕΝΙΖΑ συνεργάζεται με όλα τα διαφορετικά μέρη στον τομέα αυτό, κοινωνία των πολιτών, πολίτες, ε, κλάδο, ιδιωτικό τομέα, αλλά και η διεθνή συνεργασία είναι πολύ σημαντική, ιδίω σήμερα, όπου βλέπουμε για παράδειγμα στον ΟΗΕ ότι έχουμε δύο παράλληλες συζητήσει για το μέλλον ε, τη ασφάλεια στο διαδίκτυο. Εσείς πού εντοπίζετε το ρόλο της ΕΝΙΖΑ. Ήδη να λάβουμε υπόψη ότι είστε ένας από τους φορείς που συμπληρώνουν την ευρύτερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στον κυβερνό Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γαμών. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Σπανού για την παρουσίασή σας, πολύ ενδιαφέρουσα να μιλήσουμε για αυτά που έχουν αλλάξει ήδη, αλλά θέλω να σταθώ σε αυτά που θα αλλάξουν ε, από εδώ και πέρα. Εσείς πώς βλέπετε τη μελλοντική σχέση μεταξύ του αρμοδίου ε, κέντρου της Επιτροπής και των κρατών μελών. Θεωρείτε ότι θα υπάρξουν κάποια ζητήματα στο μέλλον, στο εγγύης μέλλον, σε ό,τι αφορά τον τομέα δραστηριοποίηση και εστίαση ε, των ε, φορέων. Μετά, τι πρέπει να κάνουμε σε επίπεδο χρηματοδότησης για να λειτουργήσουν καλά. Το κέντρο αυτό είπατε ότι θα λειτουργήσει από κοινού και με άλλους φορείς. Η Digital Europe δεν έχει κάτι αντίστοιχο. Κάποιες φορές υπάρχουν ε, συγκεκριμένα όρια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποια συγκεκριμένη εικόνα για τη χρηματοδότηση από τον τομέα που υπάρχει άλλη μεταξύ του στρατιωτικού και μη στρατιωτικού σκέλους ε, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και μετά για την συγχρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη. Το Competence Center δεν απαριθμίζεται στη συμφωνία ως εταιρική σχέση. Η Επιτροπή λοιπόν πώς θεωρεί ότι θα πρέπει να διαμορφωθούν οι αρμοδιότητες ε, αυτού του κέντρου σε σχέση με τη χρηματοδότηση. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καρβάλιο. Ευχαριστώ. Εξαιρετική η παρουσίαση. Αρχικά, πράγματι, είναι πολύ σημαντική η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για την Ευρώπη και λαμβάνει όλον και μεγαλύτερη αξία. Στο παρελθόν όμως, είχαμε κάποια προβλήματα με τα κτίρια. Έχετε δύο γραφεία στην Αθήνα και στο Ηράκλειο. Έχει ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα πλέον για να μπορέσετε να επιτελέσετε το έργο σας. Δεύτερον, αναφέρθηκε προηγουμένως από τους συναδέλφους για το 5G όπου τίθεται ζήτημα τεχνολογικής ηγεσίας. Ποιο είναι ο ρόλος του Ίζα λοιπόν, ούτω ώστε να μην ε, μείνουμε πίσω ως Ευρώπη. Και τέλο, ο αντιπρόεδρο Ανσίπ και ο Πρόεδρος Γιούγκερ ζήτησαν επιστημονική γνωμοδότηση για το μέλλον της ασφάλειας στην κυβερνοχώρο ε, στην ανεξάρτητη ομάδα υψηλού επίπεδου και εκεί λοιπόν, σε αυτή την επιστημονική γνωμοδότηση, τονίζεται ο κίνδυνος ε, μεμονωμένη προσέγγισης που δημιουργεί τροτά σημεία σε διάφορους ε, επιμέρους ε, κλάδους. Γιατί ο κάθε κλάδος διαμορφώνει εξεχωριστά μία δομή ανταπόκρισης. Υπάρχει λοιπόν κίνδυνος να μην υπάρχει διαλειτουργικότητα και έτσι να είναι πιο τροτό το σύστημα συνολικά. Πώς εσείς αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Αναφερθήκατε στην, στις γραμμέ γραμμές για την ασφάλεια, αλλά μετά και για τη σχετική νομοθετική πράξη υπάρχει και μία αντίδραση στην ιδέα εισαγωγής υποχρεωτικών ελάχιστων κατευθυντήριων γραμμών για την ασφάλεια. Βλέπουμε όμως ότι η αγορά είναι γεμάτη από μία ασφαλή προϊόντα και όλα είναι και περισσότερα συνδέονται με το διαδίκτυο. Εσείς βλέπετε πώς θα μπορούσαμε σύντομα να εισαγάγουμε τουλάχιστον αυτές τις ελάχιστες ε, προϋποθέσεις ε, για ένα ε, καθεστώς ή σύστημα πιστοποίησης. Ευχαριστώ. Κουμπίλιους. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι νέο μέλος ε, επειδή προχωρούμε από την εθνική πολιτική σκηνή, μπορώ να τα βλέπω λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Τι είδου εντολή έχετε για να παρακολουθείτε την κατάσταση σε εθνικό επίπεδο και τι είδους ε, μέσα χρησιμοποιείτε για να απαιτήσετε ανάληψη δράσης από τις εθνικές κυβερνήσεις αν δείτε ότι ε, υπολείπονται γιατί βλέπω πολλές αναλογίε και ομοιότητες ε, με τον τραπεζικό κλάδο, για παράδειγμα. Μάθαμε πολλά από την πρόσφατη ε, παγκόσμια κρίση. Είδαμε ότι κάποιες χώρες ε, παρουσίαζαν αδυναμίες, αλλά τελικά τι εξεπλήγησαν, όλοι υποφέραμε. Υπάρχουν ομοιότητες και με την ασφάλεια στην κυβερνοχώρο. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών, αλλά προχωράμε πλέον και στην εποπτεία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Διαμπάλοβα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Είναι πολλά τα ζητήματα επιτάπητο ε, που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Τώρα, εγώ θα ήθελα να θέσω ευρύτερα ζητήματα. Ξέρουμε ότι τα δεδομένα όλο και περισσότερο ε, κατευθύνουν την αγορά ποια θα είναι η συμβολή της ΕΝΗΣΑ σε ό,τι αφορά την προστασία δεδομένων και ιδιαίτερα σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει κάποιο σχεδιασμός για το μέλλον και μετά πιο συγκεκριμένα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάποιες φορές ε, μιλούμε για την κυβερνοασφάλεια ε, από εθνικής ε, σκοπιάς, αλλά ολοένα και περισσότερες επιθέσεις τρέφονται κατά μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τα καταφέρνουν γιατί είναι μικρές αυτές οι επιχειρήσεις, έχουν περιορισμένους πόρους, υπάρχει και, και πιθανότητα ανθρωπίνου σφάλματος. Επομένως, η Επιτροπή εξετάζει τον δεχόμενο καταρτήσεων, ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και το καθεξής. Και πάλι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, η δημιουργία ενός συστήματος διαπίστευσης ε, για την ασφάλιση του κυβερνοχώρου θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κάτι που εμείς δεν θέλουμε ποτέ. Επομένω, θα μπορούσε αυτό να υλοποιηθεί με έναν φιλικό προς τις επιχειρήσεις τρόπο. Ευχαριστώ. Ωραία, κύριε Σπυράκη. Ευχαριστώ. Χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ. Δύο ερωτήσεις μόνο γιατί έχουν ακουστεί και προηγουμένως. Είναι σημαντικό για μας να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείτε και συνεργάζεστε με τα κρατη τι είδου εργαλεία χρησιμοποιείτε για αυτή τη συνεργασία και τι είδου ενημέρωση έχετε τελικά και για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, στο δημόσιο τομέα, αλλά και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Δεύτερον, το θέμα τη χρηματοδότησης. Ποια είναι η γνώμη σας, τι είδους χρηματοδοτική υποστήριξη χρειάζεστε. Θα χρειαζόσασταν και εθνική χρηματοδότηση η χρηματοδότηση από υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ευχαριστώ, κυρία Βάης. Thank you. Ευχαριστώ. Ιδιαίτερα καθησυχαστική σχεδόν θα έλεγα ε, παρουσίαση για το σύστημα της ασφάλειας ε, στον κυβερνοχώρο και το πώς λειτουργεί προς το παρόν. Όμως πάντα υπάρχει αυτό το μικρό αλλά. Εγώ είμαι νέο μέλος και αν πρέπει να γυρίσω στη Δανία, στη χώρα καταγωγής μου, και να διασφαλίσω και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και χαίρομαι που αναφέρθηκε προηγουμένως αλλά και να διασκεδάσω τις ανησυχίες των συναδέλφων σε ό,τι αφορά τις, ε, την ασφάλεια, ιδίως σε σχέση με την δημόσια υγεία. Θα ήθελα να μας πείτε ποιους στόχους θα πρέπει να θέσουμε εμείς εδώ για το μέλλον. Γιατί από την παρουσίασή μας σας θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι όλα βαίνουν καλώς και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ξέρω ότι είναι μία εκλεκευμένη προσέγγιση, αλλά και εγώ ως πολιτικός θα πρέπει και εγώ να ξέρω ακριβώς ε, τι συμβαίνει και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Αν μπορείτε λοιπόν να μας παρουσιάσετε και αυτή την ε, άποψη. Και συμφωνώ με τη συνάδελφο που είπε χρειάζεται περισσότερα χρήματα, αλλά για ποιο σκοπό ακριβώς. Ευχαριστώ. Ε, thank uh, Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίως ε, για την δουλειά που κάνετε σε σχέση με την επιστοποίηση και με τον ε, μας ε, εξασφαλίζετε να μας ε, προστατεύετε κάθε μέρα ε, στον χώρο της κυβερνοασφάλειας. Ε, η δική σας η άποψη, ποια είναι η άποψή σας για τη σχέση ανάμεσα στην κυβερνοασφάλεια και την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση. Υπάρχουν όλο και περισσότερες κυβερνοαπειλές από μη δημοκρατικά καθεστώτα. Αναφερθήκατε σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις, αλλά Ποιε είναι όχι μόνο οι αμυντικές αλλά και οι επιθετικές ε, ικανότητες ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μήπω τα έχουμε αφήσει αυτά όλα στο κέντρο αριστείας του ΝΑΤΟ το θέμα της κυβερνοασφάλειας και τελευταία ερώτηση ο κύριος Φλέγκο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε ε, ακούσαμε πάρα πολλές ερωτήσεις, πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα και είμαι ευτυχής ε, που συμφωνούμε ε, πολύ σημαντική δουλειά της ΕΝΙΖΑ. Στο μέλλον θα αντιμετωπίσουμε παρεμφερείς απειλές ε, και αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία με τα κράτη-μέλη μέσα από την εκπαίδευση, την κατάρταση και την διαχείριση των κρίσεων. Επίσης ε, πρέπει να ε, δραστηριοποιηθούμε προς την κατεύθυνση του να έρθουμε σε επαφή γενικότερα με τους πολίτες, τα πανεπιστήμια, τους φοιτητές. Η δική μου πρόταση είναι η εξής έχουμε χρήματα να διαθέσουμε, άρα θα υπάρχουν και περισσότεροι υπάλληλοι στο φορέα, αλλά πρέπει να επενδύσουμε και στο μάρκετινγκ, στο να υπάρξει ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις υπάρχουσες απειλές. Και η ερώτηση είναι η εξής. Προχωράμε ε, προς το ε, σύστημα Internet of Things. Εσείς ε, τι μπορείτε να μας πείτε, τι κάνει ο φορέας σας και πώς μπορεί να αυξηθεί η ασφάλεια, γιατί το Internet of Things ε, αναμφίβολα είναι το μέλλον. Ο κύριος Φίστοφ. Πολύ συντόμα. Γνωρίζετε ότι τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε πολύ σοβαρά προβλήματα ε, στην, ό,τι αφορά την κυβερνοασφάλεια στη Βουλγαρία. Είχαμε διαρροές ε, του εμπορικού Μητρώου και την περασμένη εβδομάδα είχαμε πολύ σημαντική διαρροή προσωπικών δεδομένων, ε, πάνω από 5 εκατομμυρίων ε, πολιτών. Εσείς ήρθατε σε επαφή με τις βουλγαρικές αρχές και έχετε προχωρήσει σε συστάσεις. Τώρα πραγματικά τελευταίο στον κατάλογό μου, ο κύριος Χάισελ. Ε, θα ήθελα να επανέλθω στο δίκτυο 5G. Θα μεταδίδονται περισσότερα δεδομένα, μεγαλύτερο όγκος και ίσως 100 ε, φορές ε, πιο γρήγορα από ότι τώρα με το σύστημα 4G και ίσως ε, να υπάρξουν και περισσότερες ε, προκλήσεις ε, στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Ξέρουμε ότι γίνεται αναφορά σχετικά με τις εξελίξεις, την, το παιχνίδι ισχύω ανάμεσα στις ΗΠΑ, την Κίνα, ποιος θα πρωτοπαρουσιάσει το 5 αλλά Υπάρχουν πολλές αναπάντητες ερωτήσεις σχετικά με το τι είναι το 5G. Είναι πραγματικά ασφαλές. Είμαστε σε θέση να ε, μεγιστοποιήσουμε ε, τον όγκο των δεδομένων που να μεταδίδονται με ασφαλή τρόπο. Γνωρίζω πολύ καλά ότι θα χρειαστούμε πολύ χρόνο, ίσως ε, εκατοντάδες δισεκατομμυρίων που πρέπει να επενδυθούν, που ακριβώς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν θέλει και κάποιος άλλος ε, να λάβει το λόγο. Νομίζω οι ερωτήσεις που έγιναν ήταν ε, πραγματικά στοχευμένες και δείχνουν ότι το ξέρετε, το κατέχετε το θέμα και η Επιτροπή Βιομηχανίας ε, ε, θα βρίσκεται πάντα στην αιχμή του δόρατος για την ΕΝΙΖΑ αλλά και για το θέμα της ε, κυβερνοασφάλειας. Τώρα, σας καλώ αν θέλετε να τοποθετηθείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ στοχευμένες ερωτήσεις σας. Να σας πω το εξής. Εγώ δεν είμαι διευθύντρια της ΕΝΙΖΑ. Νομίζω δεν το κατέστησα σαφές. Είμαι διευθύντρια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρμόδια για την κυβερνοασφάλεια. Και ένα κομμάτι της ευθύνη μου είναι η εφαρμογή του κανονισμού για την ΕΝΙΖΑ, για τον φορέα ΕΝΙΖΑ. Συνεργαζόμαστε με το φορέα αυτό, ε, είμαστε αρμόδιοι για τους πόρους της ε, ΕΝΙΖΑ του Φορένιζα και πάρα πολλά άλλα, αλλά ε, πάρα πολλά θέματα που αφορούν στον Ενίζα. Θα προσπαθήσω να τα απαντήσω γιατί συνεργαζόμαστε, αλλά ο ρόλος μου ε, δεν είναι όπως σας είπα στον Ενίζα. Εγώ εργάζομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, φοβάμαι ότι δεν ήταν σαφές αυτό. Σας ευχαριστώ κυρία Νίμπλα για την υποστήριξή σας και για την πράξη σχετικά με την κυβερνοασφάλεια. Ε, πολύ σωστά είπατε ότι όλα αυτά τα θέματα, η κυβερνοασφάλεια συζητιέται πάρα πολύ σήμερα ανά τον κόσμο. Όταν λοιπόν πρόκειται για την ασφάλεια του δικτύου 5G, ε, γιατί αυτό εμπίπτει στις αρμοδιότητές μου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του έτους ε, ενέκρινε μία σύσταση προς τα κράτη-μέλη για το πώς ε, να διασφαλίσουν την ασφάλεια του δικτύου 5G. Γιατί βρισκόμαστε ε, στην διαδικασία των διαγωνισμών ε, για το σύστημα 5G. Η σύσταση λοιπόν προβλέπει μία προσέγγιση, εναρμονισμένη προσέγγιση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου πρώτα θα κάνουμε τον, την αξιολόγηση κινδύνων, ε, μετά, τι γίνεται σε σχέση με τις απειλές και κατόπιν υποτίθεται θα προτείνουμε εργαλεία για να ε, αμβληνθούν αυτοί οι κίνδυνοι. Αυτή η σύσταση υιοθετήθηκε το Μάρτιο του 2019 και τα κράτη-μέλη συνεργάστηκαν σε μια πλατφόρμα συνεργασίας είναι λοιπόν εδώ ένα παράδειγμα του τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτήν την ομάδα έχουμε τα 28 κράτη-μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον φορέα ΕΝΙΖΑ που χαράσουν πολιτική ε, και έχει ξεκινήσει η δουλειά ε, για την αξιολόγηση κινδύνων. Τώρα, ε, καταληκτική ημερομηνία για να καταθέσουν τα μέλη της προτάσεις τους ήταν η 5η Ιουλίου ε, μπορώ αν θέλετε να σας στόλω, στείλω το υλικό γιατί βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα η Επιτροπή και η ΕΝΙΣΑ ε, καλούνται να αξιολογήσουν αυτούς τους κινδύνους και μετά να καταθέσουν μία έκθεση με τα συμπεράσματά τους. Αυτή είναι αξιολόγηση κινδύνων όχι μόνο τεχνικών αλλά και πολιτικών. Η Ενίζα επίσης ε, έχει αναλάβει να κάνει ένα από τα πράγματα που γνωρίζει καλά, δηλαδή να παρουσιάσει ένα τοπίο απειλών για το σύστημα Και η Ενίζα είναι ο μόνος φορέας ε, που Ήδη το 2015 είχε σκιαγραφίσει αυτό το τοπίο, άρα δηλαδή τώρα πιο συγκεκριμένα θα αρχίσουμε να εξετάζουμε θέματα 5G. Και πριν από το τέλος του έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποτίθεται θα προτείνει μία σειρά αμβλυντικών ε, μέτρων για να μειωθούν οι κίνδυνοι. Όσον αφορά τώρα την επιστοποίηση, γιατί ετέθη αυτό το ερώτημα, η σύσταση αναφέρει ότι την ημέρα που θα έχουμε μία πιστοποίηση για το 5G στην Ευρώπη, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να το κάνουν ε, ε, υποχρεωτικό. Άρα δηλαδή αυτό ήδη είναι ένα ε, αμπλυντικό μέτρο. Για την ασφάλεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει και τις επιπτώσεις που θα υπάρχουν στην υγεία από το δίκτυο 5G. Έχουμε δηλαδή και μία ξεχωριστή επιστημονική μελέτη που γίνεται για το θέμα αυτό. Υπάρχει βέβαια και μία διασύνδεση με την πιστοποίηση. Όσον αφορά τώρα, εσείς ε, συγχαρήκατε την Ενίζα για ένα έγγραφο για την ε, ε, πληροφορική της, ε, την πολιτική. Ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Δεν αφορά εμάς. Η Ενίζα δημοσίευσε αυτό το έγγραφο. Όσον αφορά στην διεθνή συνεργασία. Αυτό είναι κάτι που νομίζω δεν το έχουμε συζητήσει ικανοποιητικά, δηλαδή έχουμε συγκεκριμένο διάλογο με όλους τους βασικούς μας εταίρους και αυτά γίνονται σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, έχουμε υπηρεσίες για την κυβερνοασφάλεια, συνεργάζονται και είναι πολύ σημαντικό για τη χάραξη πολιτικής, ε, για να υπάρχει μια κοινή πολιτική, ε, εξαρτώμεθα πάρα πολύ από το διάλογο για κυβερνοασφάλεια. Η ΕΝΙΖΑ μπορεί να συνεργαστεί με ομολόγους, αυτό προβλέπεται στην σχετική πράξη. Αλλά και πάλι είναι θέμα κατανομής των πόρων. Θα ήθελα τώρα να περάσω από τη σχέση ανάμεσα στην ΕΝΙΣΑ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας να περάσω στο δίκτυο γιατί άκουσα ότι αυτό φύγει και προηγουμένως στη συζήτηση που είχατε για τον προϋπολογισμό. Η ΕΝΙΖΑ είναι ένας αποκεντρωμένος οργανισμός ε, που στόχο έχει να βοηθήσει τα κράτη-μέλη στις υποδομές για την κυβερνοασφάλεια. Να γνωρίζουν τα κράτη-μέλη πώς αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους επιθέσεις. Ε, άρα δηλαδή ε, βρίσκεται και στο επίπεδο στην πλευρά των γνώσεων αλλά και των επιχειρήσεων. Όσον αφορά την ε, καινοτομία, εμείς έχουμε χρησιμοποιήσει διάφορα μέτρα από το πρόγραμμα ε, Ορίζοντας, ε, αυτό αναφέρθηκε και προηγουμένως, ε, για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο η Κομισιόν έχει δύο εργαλεία όπου η κυβερνοασφάλεια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Το πρώτο εργαλείο είναι Horizon Europe. Εκεί η κυβερνοασφάλεια γίνεται βικίμνια για την κυβερνοασφάλεια, αλλά έχουμε και το Euro Ευρωψηφιακό πρόγραμμα Εκεί εξετάζεται και η κυβερνοασφάλεια ε, ως ένας τομέας που πρέπει να παίξει ρόλο. Ο, ρόλο, ο λόγος γιατί προτείνουμε να συσταθεί αυτό το κέντρο είναι και διότι θέλουμε να υπάρχουν γνώσεις ε, που θα ε, καλύπτουν τις οικονομικές δυνατότητες. Έχουμε επενδύσει αρκετά στην έρευνα, αλλά Δυστυχώ, αυτά τα προγράμματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, αλλά τη στιγμή που ολοκληρώνονται δεν φτάνουν στην αγορά. Ε, και κατόπιν γίνονται πάντα από τους ίδιους φορείς, άρα θέλουμε όποιος ε, ε, έχει αριστεία σε αυτό τον τομέα να την προσφέρει. Η Ήτρε εδώ μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Είχαμε δύο τριμερείς διαλόγους και εξακολουθούμε τις συζητήσεις στο Συμβούλιο για τον τρίτο διμερή διάλογο, όποτε θα είστε έτοιμοι βέβαια, και προτείνουμε ένα σύστημα τριών επιπέδων. Προτείνουμε πρώτα απ' όλα να ε, συγκεντρωθούν όλα τα κέντρα κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη. Πέρυσι κάναμε μία μελέτη και εντοπίσουμε 650 τέτοια κέντρα στην Ευρώπη από μικρά εργαστήρια μέχρι μεγάλους ε, ερευνητικούς οργανισμούς. Η ιδέα λοιπόν είναι να υπάρχει μια ένωση που σε όλα τα κράτη-μέλη θα διοικείται από ένα κέντρο κυβερνοασφάλειας που θα χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Και έτσι τα κράτη-μέλη που δεν θα έχουν την ε, δυνατότητα ε, να προχωρήσουν, γιατί ετέθη αυτό το ερώτημα, η όλη ιδέα είναι ε, να δοθούν χρήματα και σε μη κράτη-μέλη. Και στο δεύτερο επίπεδο έχουμε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αρμοδιότητας, Ικανότητας που θα τα ε, συντονίζει όλα αυτά και θα αποφασιστεί εκεί κατά πόσον θα γίνει ε, έρευνα και πού θα γίνουν και οι επενδύσεις. Πρόκειται για μια αρκετά καινοτόμα προσέγγιση, αλλά για να σας απαντήσω και για τη στρατηγική αυτονομία, πρόκειται ακριβώς γι' αυτό ε, το να συγκεντρώσουμε πόρους και να αποφασίσουμε ε, τι θα ε, δαπανίσουμε, τι θα επενδύσουμε σε αυτόν τον τομέα όπου χρειαζόμαστε λύσεις και μέσα από το ευρωψηφιακό πρόγραμμα μπορούμε να πετύχουμε λύσεις. Με ρωτήσατε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το κέντρο ε, δεξιοτήτων, Competence Center, δυστυχώς δεν έχει επαρκή χρηματοδότηση, γιατί ε, δεν έχει να κάνει σχέση με τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Μέσα από αυτό όμως πολλά κρατημέλη έχουν μία δική τους φωνή. Πρόκειται για μία περίπλοκη πρόταση, μία πρόταση όμως που μπορεί να σημάνει τη διαφορά. Μου κάνατε και την ερώτηση για τη συγχρηματοδότηση. Αυτό είναι ένα θέμα που το συζητάμε αυτή τη στιγμή με τα κράτη-μέλη. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για τα κράτη-μέλη. Οι παράμετροι ε, του πώς ε, λαμβάνονται οι αποφάσεις για κάθε πρόγραμμα. Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω, γιατί ε, η εντολή είναι δικό τους θέμα. Ακριβώς αυτό συζητάμε τώρα με τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο έχει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Είχατε εδώ την Φιλανδική Προεδρία και ξέρω ότι αυτό είναι μία από τις προτεραιότητές σας. Όσον αφορά τώρα την πιστοποίηση ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τώρα ε, δεν μπορούν να επιτύχουν εύκολα την πιστοποίηση γιατί αυτό είναι πάρα πολύ δαπανηρό. Έχουμε ένα σύστημα αμοιβαία αναγνώρισης το οποίο κοστίζει πάρα πολύ και είναι πολύ δύσκολο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να καλύψουν το κόστος. Ε, με ένα ευρωπαϊκό σύστημα και με μία προσέγγιση της μονοπευθυντικής στηρίδας θα υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες να πάει κανείς σε ένα εθνικό εργαστήριο για να υποκτήσει ένα πιστοποιητικό. Θα έχουμε την ευκαιρία με ένα πιστοποιητικό σε μια χώρα να το εφαρμόσουμε σε όλη την Ένωση. Αν δείτε την ε, μελέτη αντικτύπου για την πρόταση πιστοποίησης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσει ήταν ε, ο βασικό λόγο τη πρότασή μα, γιατί η μικρομεσαία επιχειρήση πρέπει να πάει να πληρώσει σε κάθε χώρα όπου αναγνωρίζει το πιστοποιητικό. Αυτή είναι η προσέγγιση του One Stop Shop. Τώρα, μιλήστε για το ίντερνετ των πραγμάτων, προς τα που θα πάμε. Με βάση το νόμο για την ασφάλεια πρέπει να έχουμε ένα ετήσιο πρόγραμμα εργασία που αποφασίζει τις προτεραιότητες της πιστοποίησης. Σήμερα, η πόροι για την πιστοποίηση τη Ένωσης που τι θα σας πω ε, τέσσερις πέντε άνθρωποι είναι Υπάρχει ένα συνάδελφο από την Ενίζα εκεί. Ίσως στο τέλος του έτους να διπλασιαστούν. Αλλά πάλι για πολύ λίγους ανθρώπους μιλάμε. Άρα η προσέγγιση πρέπει να είναι step by step. Μετά, να αναπτύξουμε πρότυπα. Τα πρότυπα θέλουν χρόνο. Πρέπει να δοθούν προτεραιότητες και από πλευρά των οργανώσεων. Αλλά θεωρούμε ότι υπάρχει μια ευκαιρία στον τομέα των, του ίντερνετ των πραγμάτων. Μπορώ να σας πω την εμπειρία που είχαμε τα κράτη-μέλη. Συναντηθήκαμε άτυπα με την ομάδα πιστοποίησης κυβερνοασφάλεια των κρατών μελών που είναι άτυπη και δημιουργήθηκε από το νόμο για την κυβερνοασφάλεια στι 12 Ιουλίου. Τέσσερα κράτη-μέλη ετοιμάζουν αυτή τη στιγμή πιστοποίηση σε εθνικό επίπεδο για το ίντερνετ των πραγμάτων. Αυτό δίνει αέρα στο, στην πρόταση για να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δυνατότητες να χρησιμοποιήσουμε και να δώσουμε προτεραιότητα. Και για όλα τα συνδεδεμένα προϊόντα. Η πιστοποίηση, δεν είναι ο μόνο τρόπο, είναι ένα τρόπο για να εξασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα που φτάνουν στην ευρωπαϊκή αγορά έχουν κάποια εξασφάλιση, ότι έχουν δοκιμασιστεί, ότι έχουν αξιολογηθεί. Αυτό είναι ένα τρόπο να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Το, ε, θέμα. το ίδιο θέμα και με το 5G, με τα 5G. Πιστεύουμε ότι θέλουμε να ξεκινήσουμε την πιστοποίηση για το 5G. Έχουμε προβλήματα λόγω των ότι είναι, πρέπει να είναι πρότυπα ISO, αλλά και εδώ πρέπει να δώσουμε έμφαση. Τώρα, κρίσιμες υποδομές. Όταν συζητούσαμε τον νόμο είχαμε μεγάλη κουβέντα για τις κρίσιμες υποδομές που είναι βασικό στοιχείο της, της οδηγίας NIS που καλύπτει και το, και το ερώτημα τι θα τους πείτε όταν γυρίσετε πίσω. Ε, στην πρώτη παρουσίασή μου μίλησα για την ΕΝΙΖΑ. Τώρα μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω και για άλλα πράγματα. Η οδηγία ΙΕΝΕΣ NIS ε, επιβάλλει υποχρεώσει σε όλους τους χειριστέ ε, κρίσιμων υποδομών, νοσοκομεία, τράπεζε, μεταφορικές επιχειρήσεις να τηρούν, να πληρούν απαιτήσει ασφάλεια, αλλά δεν ορίζει τι είναι αυτές οι απαιτήσει ασφάλεια. ελπίζουμε ότι το πλαίσιο πιστοποίηση θα οδηγήσει τις επιχειρήσεις αυτές να ζητήσουν πιστοποίηση των υπηρεσιών για να δείξουν ότι πληρούν υψηλές απαιτήσει ασφάλειας. Αλλά υπάρχει τόσο πάνω ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο με αυτές τις υποχρεώσεις που, ξεκίνησαν, που ξεκίνησε πέρσι. Θα, του, θα το δούμε πώς προχωράει. Υπάρχει υποχρέωση των κρατών μελών να, να ενημερώνουν την Κομισιόν κάθε χρόνο για το αν αναφέρουν ε, επεισόδια ή φορείς, είναι και αυτό υποχρέωση. Το 2021 σε δύο χρόνια δηλαδή πρέπει να το ξαναδούμε και το τομέα των κρίσιμων υποδομών είναι ένα τομέα που θα δούμε κατά πάση αλλά αυτό εξαρτάται και από τι κατευθύνσει πολιτική που θα μα δοθούν και η οριστήσα νέα πρόεδρο έχει αναφέρει ήδη ότι η κυβερνοασφάλεια είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων τη. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι. Τι χρειάζεται η ΕΝΙΖΑ και ποια είναι η σχέση της ΕΝΙΖΑ με όλους τους άλλους θεσμούς. Τώρα, είπαμε, η ΕΝΙΖΑ έχει μικρό προπολογισμό. Με τη βοήθεια του, των συνομοθετών ελπίζουμε να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Μικρό θα μείνει όμως, ο, μικρός θα Όταν δημιουργηθεί πιστεύουμε το κέντρο δεξιοτήτων θα μπορέσει να δουλέψει και με αυτό το πλαίσιο. Αυτό τη στιγμή δεν έχει δυνατότητα. Πέραν των συζητήσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς δεν έχει άλλο θεσμικό ρόλο συνεργασίας με την κοινότητα της κυβερνοασφάλειας. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτό θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων Μα ζητήθηκε να ξεκαθαρίσουμε τα καθήκοντα αυτά και ελπίζω ότι ο τελικό, στο τελικό κανονισμό θα συμβεί κάτι τέτοιο. Άρα η ΕΝΙΖΑ χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη, αλλά αυτό που χρειάζεται τώρα περισσότερο είναι τα, οι δεξιότητε, τα προσόντα. Και η Ευρώπη και η Αμερική, στην Ευρώπη τουλάχιστον όπως και στην Αμερική, θέλουμε μέχρι το 2025 350.000 ειδικού σε θέματα πληροφορικής το λένε οι μελέτες. Είναι σημαντικό λοιπόν να αποκτήσει τις δεξιότητές της η ΕΝΙΖΑ στις επαφές με τα κρατημέλη αν θέλει να γίνει ένα κέντρο αριστείας. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που τα χρήματα δεν μπορούν να τα αγοράσουν. Μπορεί να τα αγοράσει, ε, να τα δημιουργήσει συνεργασία. Τελευταία ερώτηση. Το πώς μετράς τι είναι καλύτερο και τι είναι χειρότερο του κανόνε στην κυβερνοασφάλεια και πού είναι ο ρόλο τη ΕΝΙΖΑ εκεί. Αυτό προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την οδηγία NIS. Ήταν, η NIS ήταν ο πρώτος ε, νόμο για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη που έχει και στρατηγική και μονάδα ανταπόκρισης και αυτή την εθελούσια ε, ομάδα συνεργασίας που ήταν, το είδα πολύ θετικά τα κράτη-μέλη. Ο ρόλο ενίζει να βοηθήσει τα κράτη-μέλη που δεν έχουν την ικανότητα να την στήσουν. Μιλώντας με αυτούς που την έχουν και με λίγη βοήθεια ακόμα. Τα κράτη-μέλη όμως έχουν υποχρέωση με βάση την οδηγία να ενισχύσουν την ικανότητά τους και εμείς να τους βοηθήσουμε. Τελευταία ερώτηση για τη Βουλγαρία. Ξέρετε ότι η Επίτροπος κυρία Γκάμπρελ την ξέρει καλά τη χώρα αυτή και αμέσως ε, ε αναλάβαμε δράση, ήταν πολύ σοβαρή παραβίαση ασφάλειας, ήρθαμε σε επαφή με τις αρχές, το δίκτυο των ομάδων ε, ανταπόκρισης ε, ξεκίνησε να λειτουργεί. Γι' αυτό πιστεύουμε, αυτό έδειξε ότι το δίκτυο βοηθάει. Δυστυχώς βέβαια τέτοιες παραβιάσεις θα συμβαίνουν όλο και συχνότερα και αυτό που θέλουμε είναι η συνεργασία να βοηθάει και τη μείωση των συμβάντων σε άλλες χώρες και την καλύτερη αντιμετώπιση τους. Σχέση με την άμυνα τώρα. Στην πρόταση για το κέντρο ικανοτήτων και το συζητήσαμε εδώ εκτεταμένα, υπάρχει δυνατότητα το κέντρο δεξιοτήτων να αναλάβει να είναι ο project manager έργων κάτω από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει μετά από έτοιμα κρατών μελών που χρηματοδοτούν το ταμείο αυτό. Υπάρχει ωστόσο σύνδεση μεταξύ συνεργειών. Υπάρχει δυνατότητα συνεργειών που το είχαμε δει ήδη το 2017. Στην ουσία μερικές φορές πρώτα δημιουργούνται οι ανάγκες στον τομέα τη άμυνα και μετά φτιάχνει την ανταπόκριση σε επίπεδο κυβέρνηση ασφάλεια. Δεν ξέρω αν δεν απάντησα σε κάποια ερώτηση πρόεδρε, αν θέλετε να ξανάρθουμε με την ομάδα μου και όποιον θέλετε για να σας μιλήσω για το τι κάνουμε και βέβαια και με την νέα επιτροπή θα έχουμε και μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε τα επόμενα πέντε χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαφέστατα αυτά που μας είπατε, που παρουσιάσατε την δουλειά της Επιτροπής. Θα περιμένουμε βέβαια θα περιμένουμε το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κινδύνου για το σύστημα 5G και τα μέτρα μείωσης κινδύνου που προβλέπονται στην αξιολόγηση κινδύνου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πάρα πολύ ε, ενδιαφέρουσα συζήτηση ε, και νομίζω ότι η συζήτηση είναι και ιδιαίτερα επίκαιρη διότι τώρα έτσι έχουμε μια γενική εικόνα για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα και είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι για την επόμενη συζήτησή μας για την ΕΝΙΖΑ, για την... τον κύριο Λεπασά ο οποίος προτείνεται... Α, εδώ είναι, νάτος. Εκεί πίσω ε, σας περιμένουμε για την ανταλλαγή απόψεων στην επόμενη συνεδρίαση μας. Αυτά για σήμερα. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. 2 και 3 Σεπτεμβρίου οι επόμενες ε, συναντήσεις μας. Αλλά μέχρι τότε εύχομαι σε όλους σας ε, ηλιόλουστες διακοπές και να επανέλθετε με γεμάτες τις μπαταρίες σας γιατί σε αυτή την επιτροπή θα έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι.